Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf alle die Καλησπέρα σας, να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω όλους όσους ήλθαν στην ώρα τους. Λέει Πρόεδρος, καλωσορίζω ε, τα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου και Ρενάτα Σε ε, Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω σήμερα. Που ήλθατε λοιπόν σήμερα στην Επιτροπή μας για να μας ε, παρουσιάσετε την έκθεση για τις υπηρεσίες οι συγητές μας είναι ο Ρίτσαρτ Τσανέσκι, ο συνάδελφος Μποτζίνσκι και συνάδελφος Λεγκούτκο που έχουν μοιράσει μεταξύ τους ε, τις εξωτερικές υπηρεσίες προκειμένου για να απαντήσουν και στα θέματα που έθιξε το ελληνικό Συνέδριο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να πάρετε το λόγο και στη συνέχεια να πάρουν το λόγο οι συγγητές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να κάνω μία εισαγωγή στην ε, ελπίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα πολύ ενδιαφέροντα υποσυστήματα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, της Ευρωπαϊκής εξωτερικής υπηρεσίες. Έχετε λοιπόν τα υλικά που χρειάζεστε στην είσοδο της αίθουσας και έχετε και την παρουσίασή μου σε έντυπη μορφή. Θα είμαι συνεχτικός και σύντομος. Να ξεκινήσω όμως από την περιπλοκότητα του υποσυστήματος των ευρωπαϊκών οργανισμών. Κοιτώντας τον προπολογισμό και ο προπολογισμό τους αναλογεί σε λιγότερο από 3% του συνολικού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού ετησίως. Διαπιστώνουμε όμως και την περιπλοκότητα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση τους οργανισμούς. Έχουμε καταμετρήσει τουλάχιστον έξι διαφορετικά μοντέλα χρηματοδότησης για τις 42 αυτούς οργανισμούς, 43 από του χρόνου. Αυτό καταδεικνύει πόσο, διαφορετικέ είναι οι... πόσο διαφορετικοί είναι οι πόροι που χρησιμοποιούν. Σε ό,τι αφορά τα διοικητικά λοιπόν έξοδα, είναι εξίσου σημαντικά ο σημαντικοί οργανισμοί όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι οι οργανισμοί 1,6 δις το χρόνο ακόμα με περισσότερα. Αλλά φυσικά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μικρό το κομμάτι αυτό. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό τώρα, είναι μόνο 17% των συνολικών υπαλλήλων και προσωρινών ε, υπαλλήλων των ευρωπαϊκών οργάνων. Θα έλεγα ότι συνολικά το προσωπικό που εργάζεται για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που είναι 600.000 άτομα αναλογεί στους δημοσίους υπαλλήλους ε, των μικρών κρατομελών όπως της Λιθουανίας. Δεν περιλαμβάνουμε όμως ε, γιατρούς και αμα, δασκάλους, δημόσιους υπαλλήλους. 50-60 Παρά το γεγονός όμως ότι μιλάμε για τόσο μικρά, για μικρούς όγκους σε σχέση με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λέω πάντα και το τονίζω και τώρα, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Να κοιτάξουμε τώρα λοιπόν την έκθεση, η δική μας έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε στις 15 Οκτωβρίου. Δύο εκθέσεις δημοσιεύθηκαν. Η συνολική έκθεση για τους ελέγχους αυτό το βιβλίο που βλέπετε, αλλά και ένα σύντομο, μια σύντομη σύνοψη των εκθέσεων, την οποία, όπως σας είπα, μπορείτε να βρείτε στην αίθουσα, στην είσοδο της αίθουσας. Εκεί θα βρείτε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Να πω ότι έχουμε τρία χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή. Καταρχάς, όπως σας είπα, δημοσιεύτηκε ένα μήνα νωρίτερα από αυτό που προδιαγράφει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό κόστισε μεγάλη προσπάθεια από το ελεγκτικό συνέδριο, αλλά και από τους οργανισμούς που συμμετείχαν, που έσπρωξαν τις ε, ιδιωτικές εταιρείε ελεγκτών. Κατά δεύτερον, τα συνολικά αποτελέσματα του ελέγχου αποτελούν μια σχετικά καινούργια κρατική και αυτό δίνει μια ευκαιρία να υπάρχει μια οριζόντια παρουσίαση των προβλήματων που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί. Θα αναφέρω μερικούς εξ αυτούς. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και στην Επιτροπή εδώ, αλλά και στο Συμβούλιο που θα παρουσιάσουμε την έκθεση την επόμενη εβδομάδα. Τρίτο χαρακτηριστικό της εκθέσης μας, της με ένα πολύ απλό και ανθρώπινο τρόπο θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Επιτέλους, ε, μιλάμε για μια ενδιαφέρουσα έκθεση για οικονομικά στοιχεία. Είναι λίγο παράδοξο, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά θα είναι πιο ενδιαφέρουσα. Έχουμε τρία κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 3 έχουμε πολλές λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά όλους τους οργανισμούς, και στη μικρή έκθεση και στην ε, εκτενή έκθεση. Στο κεφάλαιο 1 ε, έχουμε το πεδίο εφαρμογή ε, του ελέγχου του Ελεκτικού Συνεδρίου και το κεφάλαιο 2 είναι πολύ σημαντικό θεωρώ. Καλύπτει τα οριζόντια θέματα και προτείνει κάποιε δράσει οι οποίε θα πρέπει να αναλευθούν σε ό,τι αφορά το δίκτυο όλων των οργανισμών. Τα αποτελέσματα τώρα. Θα έλεγα και αυτό δεν το ακούμε συχνά από το ελληνικό συνέδριο, αλλά είναι καλά τα αποτελέσματα. Μη σα πω ότι βελτιώνονται κιόλα διαρκώ. Αυτό το τονίζω. Είναι και καλά και βελτιώνονται. Και αυτό φαίνεται και στα πορίσματα, στα συμπεράσματα. Για όλους τους οργανισμούς έχουμε ξεκάθαρη γνωμοδότηση, καθαρή γνωμοδότηση. Μόνο η ΑΖΟ πήρε ε, ειδική γνωμοδότηση, qualified opinion, για το γεγονό ότι πραγματικά ακολουθούν. Ε, υπήρχε κάποια προβλήματα από πέρυσι τα οποία συνεχίστηκαν φέτο. Τα συζήτησαμε εκτενώ άλλωστε με την Επιτροπή σα και πέρσι και νομίζω ότι ο διευθυντή του οργανισμού θα μπορέσει να τα επιλύσει στη συνέχεια. Τα οριζόντια λοιπόν αποτελέσματα. Κάναμε 100 παρατηρήσει ε, και σημειώσαμε περαιτέρω ε, πρόοδο σε ό,τι αφορά τον εναρμονισμό του συστήματος πληροφορικής. Αυτό αποτελεί αποτέλεσμα τριών ετών εργασία με το δίκτυο των οργανισμών. Και τώρα λοιπόν οι οργανισμοί χρησιμοποιούν λίγο πολύ ε, τυποποιημένα συστήματα IT. Δεν χρησιμοποιούν τα δικά του. δεν φτιάχνουν τα δικά του κάθε φορά. Τώρα, τα μειονεκτήματα σε ό,τι αφορά την διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων, εδώ αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι υπάρχουν τρία παρόμοια προβλήματα σε πολλούς οργανισμούς σε ό,τι αφορά τα ε, κριτήρια απονομής των προμηθειών που δεν είναι πάντα κατάλληλα. Ε, προβλήματα σε ό,τι αφορά τιμή ε, εκπληρώση των καθηκόντων των ε, ατόμων και σε προβλήματα σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Όλα αυτά λοιπόν τεκμηριώνονται. Τεκμηριώνονται και πραγματικά ήταν ακραίες οι συνθήκες κατά τις οποίες ελήφθησαν οι αποφάσεις. Καλούμε τους οργανισμούς ε, να περάσουν στην διαπραγμάτευση και όχι να ακολουθήσουν την ε, συνήθεια διαδικασία. Ένα πιο σημαντικό θέμα το οποίο ήθελα να θέσω για τα μέλη της Επιτροπής σας είναι το θέμα των ανθρώπινων πόρων. θα ακούσετε μία ε, έκθεση την οποία κάναμε για το προσωπικό για το 2014 σε ό,τι αφορά τη σχετική μεταρρύθμιση και είπαμε ότι αυτή η περικοπή κατά 5% κόστησε στους οργανισμούς. Αμα... Ε, έγινε όμως αυτή η περικοπή και βλέπουμε λοιπόν μία τάση αμα... Ε, αντιστάθμισης της απώλειας του μόνιμου προσωπικού με προσωρινούς απασχολήμονους, με συμβούλους και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ευαίσθητα ζητήματα, αυτό δημιουργεί καταστάσεις κινδύνου. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τις πολύ σημαντικέ ε, δράσεις των οργανισμών, όταν αναπτύσσονται τέτοια καθήκοντα σε εξωτερικούς ε, εργαζόμενους, για άτομα, σε άτομα τα οποία δεν είναι υπόλογα στον Ευρωπαίο Φορολογούμενο, σύμφωνα με το καταστατικό. Αυτό το θέμα λοιπόν το υπογραμμίζω, το επισημαίνω και νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Κάποιοι τομεί τώρα βελτίωση σε ό,τι αφορά την έκθεση, σε ό,τι αφορά το πλαίσιο συντορικού ελέγχου. Υπάρχει ένα πλαίσιο μεν, θα μπορούσε να είναι πιο ταχεία όμως η εφαρμογή στους οργανισμούς. Καταχώρηση, μάλλον ε, έξοδα καταχώρησης ε, χωρίς να αλλάξει η νομοθεσία δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση στους οργανισμούς και οι οργανισμοί μπορούν να σας πούν πιο πολλές λεπτομέρειες όταν αναγκάζονται να χτυπήσουν την πόρτα των εθνικών αρχών χωρίς ε, να ξέρουν πόσα χρήματα μπορούν να έχουν στον προπολογισμό τους. Τέλος, συστημικά παρατηρούμε ότι η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής στον προπολογισμό δεν είναι ομοιόμορφη για όλους τους ε, οργανισμούς. Έχουμε αυτοχρηματοδότηση σε κάποιους οργανισμούς και η άποψη του ελεκτικού συνεδρίου, το, το λέω ξανά, είναι ότι η διαδικασία χορήγησης απαλλογή θα πρέπει να είναι η ίδια ακόμα και για τους αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λοιπόν, να χορηγηθεί η απαλλαγή αυτή. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξη για το Άσυλο θα βρείτε λεπτομέρειες το φάκελό σα, Μπορείτε να το συζητήσετε το θέμα αυτό και με τον επικεφαλής της ε, υπηρεσία Σε ό,τι αφορά την Frontex, και εδώ έχουμε κάποιες προτεραιήσεις να κάνουμε. Να υπενθυμίσω ότι αν το πρόβλημα είναι κάτω από το 2% σε κλίμακα του προπολογισμού του οργανισμού, α, δίνουμε την γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετά επαρκέ ε, και αρκετά ουσιαστικό. Να πω επίσης σε ό,τι αφορά τα σχόλια των προηγούμενων ετών έχουν πραγματικά εφαρμοστεί και ακολουθηθεί. Πολύ ικανοποιημένοι είμαστε. Για κάποια συγκεκριμένα τώρα, για κάποιου συγκεκριμένου οργανισμού, να πω ότι υπάρχουν και κάποιε ειδικέ εκθέσει, κάποιοι ειδικοί έλεγχοι απόδοση που εξετάζουν όλε του δραστηριότητε. στη διάθεσή σα για ό,τι ερώτηση έχετε, αγαπητοί βουλευτέ, και εμεί έχουμε εδώ μέλη τη ομάδα μας αν χρειαστούν τυχόν διευκρινήσει ε, και απαντήσει στις ερωτήσει σα. Σα εύχομαι μια καλή συζήτηση και τέλο χορηγούμε την απαλλαγή σε όλου του οργανισμού που πέρασαν από έλεγχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ η Πρόεδρο. ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ε, πολύ καλή αυτή παρουσίαση και χαίρομαι ιδιαίτερω που έχω μαζί μα, ε, την κυρία Γκρέκόρεφα από την ΕΑΖΟ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μα. Σας εκτιμά ιδιαίτερα η Επιτροπή μας τον τρόπο εργασία σας και το πώς ε, προσπαθείτε να διορθώσετε τα πράγματα στον ΕΑΖΟ. Ο κύριος Λεζερή επίσης, τον οποίο επίσης γνωρίζουμε μεγάλο, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και η κυρία Κάτσο επίσης ε, σας ε, καλωσορίζω. Εσείς είστε ο υπεύθυνος για τις τρεις αυτές υπηρεσίες. Γι' αυτό θα σας δώσω παραφέρον το λόγο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τα καλά σας λόγια. Ε, παρουσιάσατε έτσι τους εκπροσώπους των οργανισμών με αυτά τα εισαγωγικά λόγια. Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη από τον Ανδρέας που είναι πρόεδρος του δικτύου. Δεν μπόρεσε να έρθει και μου ζήτησε να έρθω. Γιατί ήρθα εγώ, γιατί είμαι συμπρόεδρος του δικτύου του οργανισμού ε, και αντικαθιστώ την Ανδρέα, συγγνώμη. Και από το Μάρτιο του επόμενου έτους θα αναλάβω την Προεδρία. Και έτσι θα συνεχίσουμε και τη συνεργασία μας. Ε, θα συνεχίσετε δηλαδή να συνεργάζεστε προσωπικά με μένα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που κρατάτε στην ημερήσια διάταξή σας για να γίνει αυτή η συζήτηση για τις απαλλαγές. Φυσικά πιστεύουμε ότι αυτή η διάλογοι, αυτές οι συζητήσεις είναι πολύ σημαντικό τμήμα για την νομιμοποίηση της λειτουργίας των οργανισμών και για να μας εμπιστευτούν οι πολίτες. Χάρη στη δουλειά σας, επίσης, μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε ε, βελτιώσεις σε τομείς που έπρεπε να βελτιωθούν μαζί με το ελεγκτικό συνέδριο και εσείς μας επιβεβαιώνετε ότι όντως κινούμαστε προς τη, σωστή κατεύθυνση και αυτό είναι πολύ καλό βήμα προς τους πολίτες γιατί μπορούμε να δηλώσουμε πλέον ότι είμαστε μία εύρυθμα λειτουργούσα ε, υπηρεσία, ένας καλός οργανισμός. Ευχαριστούμε λοιπόν και για τα όσα είπε το ελεγκτικό συνεδρίο για μας. Το δίκτυο των οργανισμών ε, εκπροσωπεί 47 οργανισμούς. Εγώ μιλάω για τους οργανισμούς που ανήκουν στη δική σας αρμοδιότητα μόνο σήμερα και αυτούς εκπροσωπώ. Θα συνοψίσω κάποια από τα αποτελέσματα, σκόπευα μάλλον να συνοψίσω κάποια από τα αποτελέσματα της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά το κάνατε πολύ καλά ο προλαλής σας. Μας είπατε λοιπόν ότι τα πάμε καλά, ότι βελτιωνόμαστε και ότι λίγα είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω. Άρα θα απολαύσω τα καλά λόγια του ελεγκτικού συνεδρίου, δεν θα πω τίποτα πέραν αυτού. Θέλω να διατρέξω κάποια πράγματα γύρω από αυτά που κάνουμε και κάποιους προβληματισμούς στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις πριν ακούσω τις ερωτήσεις σας. Έχω την αίσθηση ότι ως δίκτυο έχουμε προχωρήσει, μοιραζόμαστε κάποιες υπηρεσίες. Αυτό το θέμα έχει συζητηθεί πολλές φορές εδώ, Φερρυπίν κοινέ προμήθειες, ε, κοινέ διαφημίσεις για το προσωπικό, και διάφορα άλλα στοιχεία, ε, συστήματα ανάκτησης μετά από καταστροφές και μοιραζόμαστε και κάποια συστήματα πληροφορικής με την Κομισιόν. Είναι σημαντικά βήματα αυτά, πρέπει να γίνουν, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι συνολικά υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των οργανισμών ε, και είναι πολύ περίπλοκο να επιμεριζόμαστε πολλά πολλά συστήματα. Καταρχάς, ε, είμαστε τοποθετημένοι σε διαφορετικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καλό αυτό, γιατί είμαστε κοντά στους πολίτες, αλλά αυτό μας δημιουργεί λειτουργικές δυσκολίες για να μοιραστούμε κάποιες υπηρεσίες. Έχουμε μεγάλη διακύμαση στο μέγεθος των οργανισμών, έχουμε πολύ μεγάλες και πολύ μικρές υπηρεσίες για οργανισμούς. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να μοιραστούμε πράγματα. Ε, η εντολή μας, οι συμφεροντούχοι που ενδιαφέρονται για μας και τα λοιπά και, και η αποστολή μα είναι τελείως διαφορετικές. Επίσης οι οργανισμοί είναι υποτίθεται ανεξάρτητοι και επομένως δεν θα πρέπει ένας τέτοιο επιμερισμός να δημιουργήσει προσκόμματα στην εξαρτησία μας. Παρ' όλα αυτά, παρά τα προβλήματα αυτά, προχωρήσαμε στο να μοιραστούμε κάποιες υπηρεσίες. Αυτό φαίνεται από τους δύο νέους οργανισμούς που δημιουργήθηκαν και που συμμετείχαν στη τελευταία συνεδρίασή μας πριν από κανένα μήνα, όπου εποφελήθηκαν από αυτά τα κοινά πακέτα υπηρεσιών, ας πούμε, και μπόρεσαν απλώς να εποφεληθούν, ας πούμε, χωρίς να χρειαστεί να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, τρεις θα αναφέρω, τρεις βασικές προκλήσεις. Η μία είναι η ευελιξία ευελιξία κυρίως ό,τι αφορά τις συμβάσεις που δίνουμε στο προσωπικό. Συχνά οι οργανισμοί ε, έχουν διαφορετικό φόρτο εργασίας και έχουν κάποιες, περιοχές, κάποιες εποχές του χρόνου που έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Και επομένως, συχνά όταν έχουμε τέτοια πικ στη δουλειά μας, ας πούμε, ή όταν έχουμε μακροπρόθεσμα έργα ή προγράμματα, δεν είναι δύσκολο δεν είναι εύκολο να προσαρμόσουμε αυτά τα συμβόλαια, αυτές τις συμβάσεις του προσωπικού στο φόρτο εργασίας μας. Και αυτό πρέπει να το δουλέψουμε λιγάκι. Άλλες δύο προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε φέτος και στις διαπραγματεύσεις ε, και στις συζητήσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, έτσι πολύ γενικά θα τα αναφέρω αυτά τα δύο σημεία, είναι τα εξή. Καταρχάς, υπάρχει μια προσέγγιση οργανισμός που αφορά τον κάθε οργανισμό, εξατομικευμένα. Μας αρέσει αυτό, γιατί είμαστε πολύ διαφορετικοί, συνεργαζόμαστε πολύ καλά μαζί, αλλά αυτή η διαφορά μας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν ε, μιλάμε για τον προϋπολογισμό του οργανισμού, τη χρηματοδότησή του, το πρόγραμμα εργασίας κτλ. Επομένως, αυτή η προσέγγιση ανά οργανισμό, αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση είναι πολύ σημαντική λόγω των διαφορών μας. Και το άλλο σημείο, το άλλο θέμα, το οποίο μας απασχολεί εμάς τουλάχιστον, είναι ότι ακούσαμε από πολλούς οργανισμούς ότι τους ανατίθενται επιπρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες, αλλά αυτό δεν συνοδεύεται συχνά με επιπλέον πόρους ή και προσωπικό και υπάρχει η προσδοκία ότι θα τα καταφέρουν παρόλα αυτά. Μπορούν να το κάνουν μέχρι ενό σημείου, αλλά υπάρχουν κάποια όρια όταν τα ξεπεράσουμε δεν γίνεται πια να προχωρήσουμε με νέα καθήκοντα χωρίς νέους πώς. Φτάνουμε σε ένα σημείο όπου οι επιπλέον, τα επιπλέον καθήκοντα χρειάζονται επιπλέον πόρους. Με αυτά τα εισαγωγικά λοιπόν σχόλια τελειώνω την παρουσίασή μου. Θέλω να σας πω ότι πιστεύουμε ότι το δίκτυό μας με τις κοινέ ε, υπηρεσίες μας εδώ και το γραφείο στις Βρυξέλλες μπορεί να συμμετάσχει πολύ καλά στις συζητήσεις με εσά και με τους συναδέλφους από τις άλλες επιτροπές. Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε με την εμπειρογνωμοσύνη μας, με την εμπειρία μας, στο να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τις πολιτικές σας και τις πολιτικές αυτής εδώ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε και εμείς από πλευράς μας. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή του κύριο Προσίνσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω του εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου τον εκπρόσωπο του ΕΚΑ και της ΕΑΣΟ. Προσεχογικά όσον αφορά τα σημαντικά θέματα για την ανατροπή, συγγνώμη για την απαλλαγή του έτους 18, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε 40 δύο υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ένα έργο διοικητικό και διαχειριστικό. Βοηθούν σε πολλούς τομείς. Δικαιοσύνη, υγεία, ασφάλεια, ε, για τις ε, ελευθερίες και απασχολούν 11.000 υπαλλήλους στον 5 του συνολικού προσωπικού και Έχουμε πάνω από 4 δις προϋπολογισμό για το 18. 20% αύξηση δηλαδή σχετικά την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή πάνω από 7% ε, πόσο του συνολικού προπολογισμού. Από αυτές τις 42 υπηρεσίε έχουμε 32 που είναι αποκεντρωμένες και οι οποίες περνούν από τη διαδικασία απαλλαγής του Κοινοβουλίου. Το δε συνέδριο υπέγραψε τις σχετικές ε, εκθέσεις, τις ενέκρινε για αυτές τις 42 και επιβεβαίωσε την ορθότητα των ε, αποτελεσμάτων. Το Ελληνικό Συνέδριο επίσης έδωσε το πράσινο φως για όλες τις ελληνικές υπηρεσίες. Ό,τι δηλαδή οι λογαριασμοί τους είναι όπως πρέπει και επίσης και οι συναλλαγές τους και οι χρηματοοικονομικές ροές. Όλα αυτά και επίσης όσον αφορά ε, τα έσοδα και τα έξοδα. Στην ΕΑΣΟ πάντως υπήρξαν κάποιες επιφυλάξεις. Τώρα, για να δούμε ποια είναι η μεγαλύτερη κίνδυνη. Είναι θέμα αξιοπιστίας σε σχέση με αυτούς τους λογαριασμούς. Ο κίνδυνος αμεληταίο για τις περισσότερες υπηρεσίες, αλλά όλο ένα και περισσότερες αρμοδιότητες του δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει περισσότερα, πιο περίπλοκα τα πράγματα για τις ε, υπηρεσίες. Άρα υπάρχει κίνδυνος για τον προπολογισμό αυτών των υπηρεσιών. Στον αφορά την ορθότητα, στον αφορά την νομιμότητα των εσόδων, ε, είπαμε ότι είναι μικρό ο κίνδυνο, αλλά υπάρχουν και κάποιε εξαιρεσει. για την νομιμότητα των λογαριασμών χαμηλά ε, είναι τα ρίσκα και η χρηματοδότηση γίνεται από τον γενικό προπολογισμό. Υπάρχει και σχετικό κανονισμό. τα δε έσοδα από αυτόν τον προπολογισμό εγκρίνονται από τι αρχέ του προπολογισμού ετησίω. Επίση, υπάρχει κίνδυνο όσον αφορά την νομιμότητα των εξόδων των πληρωμών των υπηρεσιών. Εκεί χαρακτηρίζεται με τρίο επίπεδο ο κίνδυνο. Υπάρχουν κάποιε διαφοροποιήσει από υπηρεσία σε υπηρεσία και να συζητήσουμε λίγο τα θέματα των εξόδων για τους διάφορους τομείς. Έχουμε πρώτα πρώτα τις δαπάνες προσωπικού. Εκεί είναι χαμηλός ο κίνδυνος. Και εκεί το μισθολόγιο το έχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχουν και οικονομικοί ελεγκτές. Τα τελευταία δε χρόνια έχουν επισημανθεί σημαντικά λάθη. Όμω πρέπει να υπάρξουν πολλοί υπάλληλοι και να προσληφθούν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οπότε τότε χαρακτηρίζεται ε, μετρίου επίπεδου ή ψηλός ο κίνδυνο για αυτές τις διαδικασίες. Όσον αφορά τα έξοδα, επίσης μετά τα διοικητικά έξοδα, διοικητικέ δαπάνε. εδώ ο κίνδυνος θεωρείται μετρίου επίπεδου. Γιατί υπάρχουν διάφορες υπηρεσίες για τις οποίες πρέπει να καταληφθούν έξοδα, πληροφορική και άλλα. Άρα υπάρχει περιπλοκότητα όσον αφορά αυτές τις διαδικασίες ε, αγοράς. ούτε υπάρχει πάντοτε η αναγκαία διαφάνεια από πλευρά των υπηρεσιών. Παραδοσιακά, το ελεγκτικό συνέδριο διατύπωνε επιφυλάξεις μετά τους ελέγχους για αυτόν τον λόγο. Επίσης, τα μισθώματα των κτηρίων είναι θέμα για αυτές τις υπηρεσίες και πολλές φορές έχουμε μετακίνηση, μετακόμιση από μία έδρα σε άλλη για αυτές τις υπηρεσίες. Οπότε ε, υπάρχει επίσης κίνδυνος όσον αφορά την υπεργολαβία προς εξωτερικούς για υπηρεσίες πληροφορικής ή σε κάποιο είδους ε, πρακτορία απασχόλησης. Και εκεί υπάρχει διπλό καθεστώ, υπάρχει κοινωτική νομοθεσία, αλλά υπάρχει εθνική νομοθεσία για αυτέ τι υπηρεσίε, αυτά τα πρακτορία. Τώρα, κατά τα λοιπά, Έχουμε είτε μεγάλο ή μικρό ρίσκο ανάλογα με την υπηρεσία όσον αφορά τις δαπάνες και γενικά ο κίνδυνος σε σχέση με τις προμήθειες και τους διαγωνισμούς ε, υπάρχει εδώ η μεταβλητή του προσωπικού όμως υπάρχουν κάποιες ενισχύσεις σε σχέση με αυτά τα λειτουργικά έξοδα και κατόπιν ελέγχων είδαμε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση Όμως θα μπορούσαν οι έλεγχοι να είναι και καλύτεροι. Έχω κάποια ερωτήματα τώρα για τις υπηρεσίες. Πρώτα πρώτα για την ΕΚΑ, την υπηρεσία για τις χημικές ουσίες. Και εν προκειμένου το ελεγκτικό συνέδριο τόνισε το εξής. Υπάρχει αυτοχρηματοδότηση και ακριβώς έχει έσοδα από κάθε εταιρεία, από κάθε φορέα που θέλει να καταχωρήσει κάποιο χημικό προϊόν. Και ασκείται εκ των υστέρων έλεγχος. Φάνηκε δε ότι θα πρέπει να προσεχθούν οι πληρωμές, τα έξοδα. Όμως δεν αναφέρονται πουθενά ακριβώς ποιες, πόσες πρέπει να είναι οι διορθώσεις για να βελτιθεί το σύστημα. Δηλαδή εδώ πέρα λαμβάνεται υπόψη η δήλωση του ετούντο αύριο θα πρέπει να είναι ακριβέστερα τα αριθμητικά στοιχεία. Γεια σου. Έχω να ρωτήσω το εξή. Τι μέτρα θα πρέπει να λάβει η υπηρεσία. Έτσι. Να μην υπάρχει πρόβλημα με την ε, έλλειψη εμπειρογνώμων από τα κρατημέλη και επίσης ε, την ανεπάρκεια του προσωπικού. Επίσης, τι κίνδυνος υπάρχει όσον αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας. Τέλος, Frontex. Ο κύριος Διευθυντής τα ξέρει γιατί έχει υπηρετήσει στο Υπουργείο Ιστορικών. Γνωριζόμαστε καλά. Αλλά τώρα και από τη θέση του Ευρωβουλευτή, υπό τη νέα μου ιδιότητα, θέλω να τον ερωτήσω κάτι. Η Άσο έχει κάποιες ε, συμβάσεις με τις ε, κάποιες συνδυόμενες χώρες, δηλαδή που είναι 171 εκατομμύρια ευρώ, 59%, 59 του προπολογισμού της για τη χρήση αυτή, και επίσης με αυτές τις χρηματοδοτικές ε, συμφωνίες καλύπτει και ανάγκες προσωπικού και κάποια στιγμή ξεκίνησε ένας έλεγχος εκ των υστέρων για να καλύπτονται όλες οι δαπάνες εκ των υστέρων σύστημα ελέγχου. Και για το 2014 λέει το Ελληνικό Συνέδριο ότι η επιβεβαίωση των δαπανών όσον αφορά το υλικό, τον εξοπλισμό από τις συνδυόμενες χώρες δεν είναι αρκετά ακριβή και επαρκής. Έτσι αυτό ισχύει λοιπόν και για αυτόν τον εκ των υστέρων ε, έλεγχο τη Frontex που δεν θεωρείται τόσο αποτελεσματικό, διότι οι πληρωμές και οι δαπάνε γίνονται για κάποια έξοδα και χωρίς παραστατικά. Ακριβώς όπως και την προηγούμενη χρονιά. Δεν έγιναν σχετικά με αυτό έλεγχοι εκ των υστέρων. Επομένω, κάποιες δαπάνε θα πρέπει να ανακριθούν μέχρι το ορθό ποσό. Οπότε θα πρέπει να μας πείτε τι να κάνουμε για να έχουμε πιο σωστούς ελέγχους και τι θα πρέπει να γίνει με τις συμφωνίες με τις ιδιόμενες χώρες και όσον αφορά αυτό τον εξοπλισμό, αυτό το υλικό που αφορά τις σχετικές δαπάνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολλές ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να δώσω στον κύριο Χάνσεν και στον κύριο Λεζουερή κατευθείαν την ε, ευκαιρία να απαντήσουν, να μας πούν πώς ε, τα βλέπουν τα πράγματα. Ξεκινάει ο κύριος Χάνσεν. Και έτσι νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσει κατευθείαν στις ε, ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Δύο θέματα έχω να θέξω σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό. Άμα των τελών και κατά δεύτερον το θέμα των μικρομεσαίων. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα το λόγο στον συνάδελφο. Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των τελών, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε σε όλους τους οργανισμούς. Έγινε μια ανεξάρτητη έρευνα για τον υπολογισμό των ε, τελών και υπολογίστηκε ότι το εύρος αυτό είναι γύρω στα 10 ε, εκατομμύρια αυτό αντιστοιχεί στους υπολογισμούς μας. Αυτό είναι λοιπόν πρόβλημα σε ό,τι αφορά το συνολικό προϋπολογισμό. Για να δούμε λοιπόν ε, ποιος ε, είναι το τέλος που θα πρέπει να υπολογιστεί στον προπολογισμό και αυτό προφανώ ε, επιβαρύνει πολύ τι καθημερινέ μα δράσει. Θα θέλαμε ένα πολύ πιο βιώσιμο τρόπο για την καθημερινή μα δράση. Αυτή η διακύμανση επίση σε ό,τι αφορά το εισόδημα από τα τέλη έχει να κάνει και με την ε, διαφοροποίηση των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να δώσω το λόγο στον συνάδελφό όμω για να απαντήσει. Καλησπέρα κύριε και κύριοι. Είμαι διευθυντή στο θέμα πόρων στην Ευρωπαϊκή υπηρεσία για τα χημικά προϊόντα σε ό,τι αφορά το θέμα της επαλήθευσης του SMU, SMU. Σε ό,τι αφορά μάλλον το, την επαλήθευση του μεγέθους της εταιρεία. έχουμε να πούμε το εξή. Επισημαίνουμε ότι το ελεκτικό συνέδριο επισημαίνει ότι έγιναν προσπάθειες για να υπάρχει ένα σύστημα εκ των υστέρων επαληθεύσης. Συμφωνούμε με την παρατηρήση του Ελεκτικού Συνεδρίου ότι το θέμα της αυτοαξιολόγησης είναι προβληματικό. Αυτές οι δηλώσει για το κάθε ε, εταιρεία δυσκολεύουν για δύο λόγου. Καταρχάς είναι πολύ περιπλοκοί κανόνε για το μέγεθο τη εταιρεία και φυσικά υπάρχει και οικονομικό κίνητρο να δηλώσει κανεί μικρότερο μέγεθο από το πραγματικό μέγεθο τη εταιρεία του. Έχουμε επαληθεύσει, έχουμε μάλλον εναρμονίσει την διαδικασία επαληθεύση. Έχουμε κάνει και κάποια εξωτερική ανάθεση τη διαδικασία αυτή προκειμένου να επιταχυνθεί το όλο θέμα και συνεχίζουμε να επαληθεύουμε τις εκκρεμίσεις υποθέσεις με ε, κάποιο κριτήριο προτεραιότητα και πάλι σκοπό μας είναι να επιταχύνουμε την όλη διαδικασία. Ωστόσο, να διευκρινίσουμε ότι για μας η διαδικασία κάθε αυτή είναι μακροσκελής, απαραίτητη και επιβαρυνή. Σε ό,τι αφορά τώρα το εισόδημα, το ελεκτικό συνέδριο σημειώνει ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο για την ανάκτηση των ε, περικοπών και σε ό,τι αφορά τα τέλη. Να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο σχετικό κανονισμό για τα τέλη δεν μα δίνει τη νομική βάθηση που χρειαζόμαστε για να άμα, λύσουμε το θέμα των ε, τελών που χρωστούνται. Θα προωθήσουμε μία διπλή προσέγγιση για την ε, ίσταξη των τελών αυτών θα καλέσουμε λοιπόν τους συμβασιούχους να συλλέξουν τα τέλη αυτά και στη συνέχεια να παραπέμφθουν τα κράτη-μέλη στις εθνικές διαδικασίες εκδίκασης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Λιζερή. το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα συνεχίσω. Θα αγγλικά. Τον εκ έλεγχο που κάνουμε, για τον εκ εκ των υστέρων έλεγχο που κάνουμε, θα σας μιλήσω για το τι κάναμε το 2018 στο Frontex. Όπως είπε και το ελεγκτικό συνέδριο, περάσαμε σε ένα σύστημα μοναδιαίων ποσών, κατά αποκοπήν ποσών, σε ό,τι αφορά τους ανθρώπινους πόρους. Δηλαδή, περάσαμε σε ένα νέο σύστημα για την αποστολή ε, συνοριοφυλάκων που δίνουμε στα κράτη-μέλη, αλλά όχι για το τεχνικό εξοπλισμό, δηλαδή τα σκάφη, τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα κτλ. Για το 2018, λοιπόν, η ανάλυση κινδύνου και η αξιολόγηση που κάναμε για τον κίνδυνο ήταν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος λάθη, παραλήψεις ή διοπιστήματα ε, αφορά, αφορούν τα νέα ε, μοναδία ποσά. Γι' αυτό ενισχύθηκαν οι εκ των υστέρων έλεγχοι για την αποστολή προσωπικού στα κράτη-μέλη. Δεν κάναμε εκ των για, την, για τον τεχνικό εξοπλισμό, γιατί δεν αλλάξαμε τους κανόνες. Φυσικά μπορεί να βελτιωθεί ο κανόνας και θα το κάνουμε στο μέλλον για τον εξοπλισμό, αλλά θέλαμε το 2018 να ε, δρομολογήσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να ελέγξουμε ποιες θα ήταν οι συνέπειες των μοναδιαίων ποσών σε ό,τι αφορά την αποστολή τεχνικού εξοπλισμού. Ξεκινήσαμε και ένα διαγωνισμό για πιλωτικά προγράμματα στα κράτη-μέλη. Όμως υπήρξε μια αύξηση του κόστους και Μάλιστα, ε, τα κράτη-μέλη αυξάνουν τις τιμές τους για την αποστολή σκαφών όταν αρχίσαμε να μιλάμε για μοναδιαία ποσά. Οπότε αποφασίσαμε να τα παρατήσουμε και να περάσουμε σε μια άλλη πολιτική ε, που αφορά και το Ευρωπαϊκό Μόνιμο Σώμα. Δηλαδή, καταρχάς θα έχουμε πιλωτικά προγράμματα για να δούμε τι θα κάνουμε τις με τα δικά μας σκάφη τα οποία θα αναβλώσουμε και να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές τιμές στην αγορά. Αν πάρουμε, ας πούμε, τα σκάφη από τα κράτη-μέλη. Οι πληρωμές πάντως ε, έγιναν με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία, τα οποία υπέγραψε η αρμόδια αρχή για την διαχείριση της συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής στα κράτη-μέλη και έχουμε τη διασφάλιση ότι αυτοί οι υπολογισμοί που κάνουν τα κράτη-μέλη παρότι ήταν ε, εθελούσιες δηλώσεις, ήταν δίκαιες και δεν παρατηρήσαμε αποκλήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Επομένως, ε, καταλήγουμε ότι υπήρχε μικρότερος κίνδυνος για τον τεχνικό εξοπλισμό ε, το 2018. Το τέλος του 2018 αναθεωρήσαμε και το σύστημα εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων για να το ενισχύσουμε αυτό το σύστημα των ελέγχων ενισχύουμε τους ε, εκ των προτέρων ελέγχους με ένα γραφείο επιθεώρησης και ελέγχου για να διαχωρίσουμε καλύτερα τους ελέγχους που γίνονται πριν πριν να δεσμευτεί ο προϋπολογισμός και από την άλλη τους εκ των υστέρων ελέγχους που είναι στα, χέρια αυτού του γραφείου επιθεώρησης και ελέγχου και που δεν είναι ποτέ ε, στη δέσμευση ε, πιστώσεων του προπολογισμού. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρικόρ, Θέλω να πάρει το λόγο και πάλι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή που μας έκανε το ελεγκτικό συνέδριο και τις ερωτήσεις του εισηγητή. Η ΕΑΖΟ το 2018 πέρασε από μια μεταβατική περίοδο. Το πρώτο εξάμεινο είχαμε το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και διορίστηκε ένας προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής. Ε, δημοσιεύτηκε και ένα σχέδιο δράσης. Και το ελεγκτικό συνέδριο παραδέχεται ότι κάναμε συγκεκριμένα πράγματα για να βελτιώσουμε τη διακυβέρνησή μας, τη διαχείρισή μας σε ό,τι αφορά το προσωπικό και την προσ... τις προσλήψεις γενικά στον ΕΑΖΟ υπήρξαν προβλήματα. Το 2018 όμως ε, οι διαδικασίες πρόσληψης έγιναν πιο διαφανείς μέσω της υιοθέτηση νέων διαδικασιών και ενισχύσαμε το προσωπικό που κάνει τις προσλήψεις. Ήταν 6 και τώρα είναι 14 τα άτομα αυτά και θα συνεχίσουμε την την ενίσχυση της ομάδας αυτής. Δηλαδή θα δώσουμε... Θα έχουμε και άλλα μέλη. 219 άτομα προσωπικό είχαμε στα τέλη του 18. 89 ε, άτομα ακόμα δεν είχαν προσληφθεί και σήμερα έχουμε 310 άτομα στα γραφεία μας. Προβλέπουμε λοιπόν για φέτος προβλέπαμε μάλλον 390 άτομα. Τουλάχιστον όμως ελπίζουμε μέχρι τα τέλη του 19 να έχουμε προσλάβει το 85% των προβλεπόμενων ανθρώπινων πόρων. Προβλέπεται αύξηση του προσωπικού μέχρι και 500 άτομα μέχρι το 2020. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να προσλαμβάνουμε με αυτό το ρυθμό στην ΕΑΖΟ. Θέλω να απαντήσω και στον εισηγητή, ο οποίος μίλησε για την έλλειψη εμπειρογνωμόνων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Ξέρετε ότι με βάση την εντολή της ΕΑΖΟ μπορούμε να βοηθήσουμε ή να στηρίξουμε τα κρατη και επιτόπου αυτή τη στιγμή έχουμε επιχειρήσει σε τέσσερα κράτη-μέλη, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη Μάλτα και στην Κύπρο, τα κράτη της πρώτης γραμμής. Με βάση την εντολή μας μπορούμε να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να μας στείλουν ή να αποσπάσουν, ας πούμε, εμπειρογνώμονας για το άσυλο και να δουλέψουν στις ομάδες ασύλου μας. Αλλά οι προσλήψεις από τα κράτη-μέλη ε, είναι πολύ λίγες. Έχουμε μόνο 13 άτομα. Είναι 3% δηλαδή των εμπειρογνωμών που δουλεύουν ε, σε αυτές τις τέσσερις χώρες. Αν τα κράτη-μέλη δεν στείλουν ή δεν αποσπάσουν εμπειρογνώμονες για το άσυλο στον οργανισμό μας, θα πρέπει να βρούμε από αλλού τους πόρους. Γι' αυτό λοιπόν η ΆΣΟ έχει, αυτές, έχει έκτακτους υπαλλήλους ε, σε αυτούς τις ε, ομάδες ασύλου. Ε, τους βρίσκουμε από παρόχους ε, υπηρεσιών και εποφελούμαστε από τους υπαλλήλους μας και από τους εμπειρογνώμονες όσους μας στέλνουν τα κράτη-μέλη. Ελπίζω τα κράτη-μέλη να θελήσουν να στείλουν περισσότερους εμπειρογνώμονες στις επιχειρήσεις μας, γιατί εμείς στηρίζουμε τα κράτη-μέλη που το έχουν ανάγκη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά προβλέπει η εντολή μας. Ξέρετε ότι η Υπηρεσία Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τμήμα του πακέτου ασύλου και θα έχουμε, υπάρχει πρόταση για μια ομάδα 500 εμπειρογνωμόνων που θα είναι στη διάσταση του ΕΑΖΟ, του οργανισμού μας. Αλλά έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα μπορεί να αποδειχθεί ότι και τα 500 άτομα δεν θα επαρκέσουν. Ähm, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκιώτες, εισηγητές τώρα. Ο συνάδελφος Νοβακόφ, πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα αρχίσω με συγχαρητήρια προς τη Γραμματεία το ελληνικό του και των υπηρεσιών, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Καταλαβαίνω τους διερμηνείς και σήμερα έχουμε τις ίδιες δυσκολίες, έχουμε μια εκατοστή σελίδα για την απαλλαγή που είναι ακατανόητες για κάποιον εκτός παιχνιδιού. Οπότε η δουλειά μας σήμερα είναι να εξηγήσουμε γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά. Uh, ε, 32 agencies. Έχουμε 32 υπηρεσίες και κάνω όλη τη δουλειά. Γι' αυτό έχουμε καλά τρόφιμα, ασφαλή τρόφιμα, ασφαλείς μεταφορές. Ένα σωρό πράγματα κάνετε και πολλές φορές φαντάζομαι σας υποτιμούν. δεν, δεν, δεν ε, φτάνει το μήνυμα στον κόσμο το, το έργο σας που είναι τόσο σημαντικό. Εκατοντάδες σελίδων το αποδεικνύουν αυτό. Και έχω εδώ μια σειρά ερωτήσεων, η πρώτη γενική ε, ύφη. Νομίζω ότι το δίκτυο μπορεί να μου απαντήσει. Η Φιλανδική Προεδρία πριν δύο μέρε, όπω ίσω θα ξέρετε, είπε ότι θα υπάρξει ένα καινούριο box, μια κατηγορία. Για τι διαπραγματεύσει που φαίνεται δύσκολος ο συμβασμό στι διαπραγματεύσει γιατί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλε ε, ε, περικοπές. Φτάνουμε το 1,06% του ΕΠ το οποίο φυσικά αυτό θίγει και τις υπηρεσίες. Άρα ταυτόχρονα Ελπίζουμε εσεί να έχετε περισσότερες αρμοδιότητε, περισσότερο προσωπικό, να έχετε λιγότερα σφάλματα και πιο μικρό προπολογισμό. Πώς το βλέπετε αυτό για την ΕΑΣΟ τώρα. Κάτι θετικό. Έχετε κάνει αυτοκριτική στα τελευταία χρόνια. Ε, πάντα βοηθούσαν οι εκτελικοί διευθυντέ, αλλά η σημερινή απόφαση είναι να κλείσουν λογαριασμοί για το 2017 όσον αφορά την ε, απαλλαγή και εμεί έχουμε χειροπιαστά στοιχεία γι' αυτό. Οπότε, ένα ε, ανατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Χρειάζεται πάντω εμπειρογνώμονε. Το θέμα είναι τι θα γίνει αφού δεν υπάρχουν προ το παρόν εθνικοί εμπειρογνώμονε. Δεν είχαμε τη βελτίωση σχετικά με πέρσι για τη Frontex τώρα. Το 2018 ήταν μεταβατική περίοδο από πολλέ ε, πλευρέ και υπάρχει ένα καινούργιο σύστημα οικονομικό εξπόστα έλεγχος για να καλύψει όλες τις δαπάνες και άλλαξε το σύστημα των ελέγχων εκ των υστέρων. Οπότε τώρα περιμένουμε τους καρπούς αυτών των νέων συστημάτων. Είχατε πρόβλημα να προσλάβετε προσωπικό, έχετε κάποιο πρόγραμμα τόσο ώστε να ελκύσετε κόσμο. Και αυτό συνδέεται και με την πρώτη μου γενικότερη ερώτηση όσον αφορά τις περικοπές για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτά, αυτά. Πάνω κάτω. Ως γενικές ερωτήσεις και πιο συγκεκριμένες. Προσιάσω και Frontex. Και πάλι σας ευχαριστούμε για όλα αυτά τα οποία κάνετε κατά κάποιο τρόπο. Η Επιτροπή μας είναι ο καλύτερος φίλος του φορολογούμενου, γι' αυτό έχουμε σκληρά ερωτήματα. Αλλά να είστε σίγουροι ότι είναι η χρηματοδότηση της υπηρεσίας των υπηρεσιών σε καλά χέρια και θα πετυχαίνουμε πολλά. Καλή αλλά σκληρή. Αυτό θέλω να σου πει με λίγα λόγια. Σκληρή τις ερωτήσεις. Η σκιώδη συζήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον συνάδελφο. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και ευχαριστούμε για τη σκληρή σα δουλειά, για όλους μας. Έχω ερωτήσει και προ τις τρει υπηρεσίες. Δεν έχω να πω γενικές πατρίσει γιατί τι έχουν πει άλλοι να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια όσο γίνεται. Έτσι κι τα ίδια ζητήματα ε, αναδύονται και εξετάζουν. Πρώτα πρώτα, υπηρεσία για τα χημικά. Συγγνώμη γιατί το έχουμε ξαναπεί, αλλά θέλω να το τονίσω. Βλέπω στο 3.7.13 τα εξή. Υπάρχει κίνδυνος ότι οι αξιόπιστες δαπάνες και μη προβλεπόμενα είσοδα θα επηρεάσουν τη λειτουργία της υπηρεσίας και την εκτέλεση του προπολισμού. Η ΕΚΑ, επομένως, λέει ότι θα πρέπει να αρχίσει επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υπάρχει κάποιο νέο μοντέλο χρηματοδότησης βιώσιμο. Και σας ερωτώ, γιατί το μοντέλο αυτό συζητήθηκε σύντομα στον προηγούμενο γύρο. Πέστε μας, τι λέτε για αυτό το σχόλιο του Ελληνικού Συνεδρίου. Και ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό το βιώσιμο μοντέλο χρηματοδότηση. Αυτό για την ε, ΕΚΑ. Θα κόψω λίγο από αυτό που θέλω να πω γιατί είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος. Ευχαριστούμε που ξαναήρθατε κύριε. Τα έχουμε ξαναπεί όταν κάναμε την ε, τελευταία έκθεση του 16 για την απαλλαγή και σας ρωτώ Α, μισό λεπτό για να δούμε πρώτα πρώτα τις συστάσεις για την ΕΚΑ το είπαμε, το είπαμε όμως αυτό που ήθελα να πω, θα το παραλείψω αλλά θα ήθελα να ξαναγυρίσω στην ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου όσον αφορά τις μετακαταστάσεις και την επιστροφή, τις επιστροφές, εάν επιτρέπετε, γιατί θέλω να μου πείτε δύο λόγια, γιατί αυτό αφορά το μέλλον. Ο, όμως, υπάρχει συντονισμός, υπάρχει συσχέτιση ΑΜΕΦ και ΕΑΣΟ, διότι στην έκθεση αυτή υπάρχουν κάποιες ε, συστάσεις για συμπληρωματικότητα και καλύτερο συντονισμό μεταξύ ΑΜΕΦ και ΕΑΣΟ. Ξέρω το είναι υπηρεσία και το είναι ταμείο. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει κάποια συνάφεια και θέλω να μου τα σχολιάσετε. Επίση, όσον αφορά του ευάλωτου μετανάστες, έχουμε κάποια στοιχεία στην έκθεση και δεν ξέρω, κάνει καμία προσπάθεια η Άσο ώστε να φροντίσει το έργο της για συλλογή δεδομένων για τους μετανάστες. Υπάρχει συντονισμό σχετικά με αυτά τα δεδομένα. Πεστε κάτι για τις ε, ελληνικές αρχές σε σχέση με αυτό. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο είδους κεντρική συλλογή στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τους ευάλωτους μετανάστες. Και τέλος για τη Frontex. μια ερώτηση και αυτό αφορά την ΝΑΜΕΦ γιατί έχουμε τις εγγραφές απαντήσεις και σας ευχαριστώ Frontex αλλά αναφέρονται τρία περιστατικά σοβαρά το 18 όσον αφορά κάποιες ε, Επιχειρήσει ε, επαναπατρισμού, επιστροφών. Η Frontex λέει, έχετε παρκείς διαδικασίε για να το κάνετε αυτό, έχετε αρκετή χρηματοδότηση και προσωπικό για να αντιμετωπίσετε τέτοια περιστατικά. Αυτό γίνεται. So, jetzt habe ich gleich drei. Μάλιστα. Έχω λοιπόν τρία άτομα από το Renew. Να ξεκινήσουμε. Ποιο θέλει να πάρει πρώτο το λόγο. Μάλιστα, οι κυρίε προηγούνται. Α, εξαριστερά. Να ξεκινήσουμε. Να σα ακούσουμε, συνάδελφοι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση και για την ε, σκληρή δουλειά. Θα προσπαθήσω και εγώ να μην ε, επαναλάβω τι ερωτήσει που ήδη ακούστηκαν από του συναδέλφου. Έχουμε κάποιε συγκεκριμένε ερωτήσει, οι οποίε ενδεχομένω να σα αφορούν όλου σα. Και ύστερα έχω μία ερώτηση να κάνω σε μία υπηρεσία συγκεκριμένα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το whistleblowing, τους πληροφοριοδότες, με χαρά σημειώνω ότι υπάρχουν ε, σε όλες τις ε, ε, υπηρεσίες ρυθμίσεις, κανόνες για τους πληροφοριοδότες και δεν έχουν παρουσιαστεί προβληματικά περιστατικά. Θα ήθελα όμω να ρωτήσω αν ε, οι υπηρεσίες σας ε, οργανώνουν ε, εκπαιδευτικά προγράμματα σε ό,τι αφορά τους πληροφοριοδότες. Γιατί έγινε έτοιμα να υπάρχει ένα εξάρτητο σώμα για παροχή τέτοιων συμβουλών, προκειμένου να βοηθηθούν οι πληροφοριοδότες να χρησιμοποιούν τις σωστές οδούς για να ενημερώνουν για ενδεχόμενες ατασταλίες οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναρωτιέμαι αν κάποιοι από τους οργανισμούς έχουν ιδρύσει τέτοια σώματα. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω πώς αντιμετωπίζετε ενδεχομένω υποθέσεις παρενόχλησης. Ξέρουμε ότι όλοι οι οργανισμοί έχουν πολιτική για την προστασία των ατόμων σε ό,τι αφορά την άσκηση ψυχολογικής ή σεξουαλικής παρενόχλησης ε, οργανώνονται όμως ε, ενημερώσεις για το προσωπικό. Πώς εφαρμόζεται λοιπόν την πολιτική αυτή. Πείτε μας λοιπόν. Nice. And the third is that, uh, Τρίτο ζήτημα. Η έκθεση αναφέρει ότι στην περίπτωση κάποιων υπηρεσιών και την ε, υπηρεσία για τα χημικά και τη Frontex αναφέρεται ότι υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από εξωτερικούς ε, παράγοντες και συμβούλους. Έχουν αναθέσει εξωτερικά λοιπόν πολλές ε, δραστηριότητες ακόμα και δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως core βασικές, κεντρικές συνάδει αυτό με το μοντέλο ή μήπω θέλετε να γίνουν αλλαγέ. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Στρουγκάριο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Συνολικά, επειδή παρακολούθησα τις εργασίες των οργανισμών και είμαι και σχεδόν συγγετρία όλος ιδιαίτερος για τις ε, υπηρεσίε στον τομέα της δικαιοσύνη και των ιστορικών ε, υποθέσεων. Ξέρω ότι αυξήθηκε σημαντικά ο φόρτο εργασία τα τελευταία χρόνια. Αυτό το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Και είμαι βέβαιη ότι έγιναν πολλές προσπάθειες σε ό,τι αφορά να... την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Ξέρω ότι έχουμε και πολλές ε, προσδοκίες και πολλές προδιαγραφές από πλευράς μας είναι σημαντικό. Και αυτό το αναφέρουμε για όλες τις εκτορικές υπηρεσίες, το ότι έχουν κάνει σημαντικά βήματα για να υπάρξει αποτροπή στο βαθμό του δυνατό τη σύγκρουση συμφερόντων και του συστήματος revolving doors. Για αυτούς λοιπόν που έχουν κανόνες για τους δημόσιους διαγωνισμούς είναι σημαντικό να συνεχίσουν να δημοσιεύονται σε ό,τι αφορά τους διαγωνισμούς, τις συμβάσεις που αντιφένται. Ξέρω ότι υπάρχουν συστάσεις για να δηλώνουν όλοι ε, ότι δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε ε, είναι η δήλωση των συμφερόντων, των οικονομικών συμφερόντων και η απουσία σύγκρουση συμφερόντων. Ίσως θα πρέπει να γίνεται αυτή η εξελόγηση από κάποιον εξωτερικό και τρίτο φορέα. Κάτι άλλο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ. Η κατάσταση που αναφέρθηκε από τους συναδέλφου σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Frontex. Για να το πούμε απλά. Το ελεκτικό συνέδριο διαπίστωσε ότι οι δαπάνες από κάποια χώρα δεν συνοδεύονταν πάντα από τιμολόγια και παρόλα αυτά αποζημιώνονταν. Πληρώνονταν τα ποσά αυτά. Και έτσι λοιπόν αυτό που αποκαλύφθηκε ότι πάνω από 300.000 ευρώ χορηγήθηκαν στην Μάλτα και στη Λιτουανία παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ποτέ λοιπόν επίσημα παραστατικά. Καταλαβαίνω ότι άλλαξαν οι διαδικασίε παρόλα αυτά. Είπατε και στην απάντησή σας ότι οι εθνικές αρχές υπέβαλαν εναλλακτικά τεκμήρια. Ωστόσο, τι ακριβώς είναι αυτά τα εναλλακτικά παραστατικά τα οποία υποβλήθηκαν. Ήταν επαρκή. Γιατί δεν είχαν διευκρινιστεί αυτά τα εναλλακτικά παραστατικά εξ αρχής. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να δαπανούμε με τον τρόπο αυτό τα χρήματα των φορολογμένων. Και σε ό,τι αφορά ευαίσθητης τομείς πολιτικής και πάλι στρέφομαι προς την Frontex, από ό,τι απαντάτε στην ΕΚΑ, είπατε ότι θα ισχύσει νέα πολιτική από τις αρχές του 2019. Δεν έχει γίνει όμως κάτι τέτοιο έως τώρα. Ή μήπως έχει γίνει. Αν έχει γίνει, να μας δώσετε πιο πολλές λεπτομέρειες. Ένα γενικό σχόλιο για την ΕΑΖΟ το 2018 ήταν ένα δύσκολο ενδιάμεσο έτος με κάποια μόνιμα ζητήματα σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, ε, κανόνες που δεν ακολουθήθηκαν. Ωστόσο, τώρα, έχουμε πλέον ε, η νέα Γενική Διεύθυνση, η οποία προσπαθεί να διορθώσει την κατάσταση. Παρακολουθώ τις προσπάθειες αυτές. Ε, δεν θα σχολιάσουμε και πάλι λοιπόν τα πράγματα που πήγαν στραβά και θέματα κατάχρησης και πόρων αλλά και διαδικασιών. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό έχω μία ερώτηση να κάνω γιατί αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πιστεύετε ότι έχει έρθει η στιγμή να προσαρμοστεί το πεδίο της εντολής των οργανώσεων και αν ναι, πώς. Και τι γίνεται σε ό,τι αφορά την εμπειρία σας από την παρακολούθηση των αρμοδιοτήτων ως τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Μπογή. Θα μιλήσω γαλλικά, πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εισηγητές για τις παρεμβάσεις τους και για τη σημαντική δουλειά που κάναν. Ευχαριστώ επίσης τους εκπροσώπους των διαφόρων οργανισμών που πήραν τον λόγο. Εγώ είμαι νέο μέλος ε, στο Κοινοβούλιο, νέος βουλευτής και είναι μια πολύτιμη στιγμή. Έχω τη δυνατότητα εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών να δω αυτή τη δουλειά που γίνεται, να την καταλάβω καλύτερα. Κοίταξα με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση και με φρίκη ανακάλυψα ότι ήταν μια περίληψη. Θα αρκεστώ την περίληψη λοιπόν. Μια γενικότερη ερώτηση Και μία ακόμα ερώτηση επί της αρχής. Όταν ρωτάμε τους οργανισμούς για, τον, για το ποσοστό εκτέλεσης του προγραμματός τους, πολλοί οργανισμοί λένε ότι κάνουν εσωτερικές ανακατατάξεις. Μερικές φορές αυτό ε, εξηγεί τις καθυστερήσεις ή δείχνει ότι γίνεται μια άλλη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Παραδείγματο χάρη, η Ευρωπαϊκή προτεραιοτητων παραδειγματος χαρη η ευρωπαικη αρχη χρηματαγορών. Μας λέει ότι σε ό,τι αφορά ε, τον κανονισμό για τα ταμεία, έχουν νέες, νέα καθήκοντα, αλλά χωρίς νέους πόρους. Και χρειάστηκε λοιπόν να ξαναβρει ε, προσωπικό, να αναθέσει ας πούμε, τα νέα καθήκοντα στο προσωπικό, εις βάρος των παλιών ας πούμε, καθηκόντων του. Αυτό δεν είναι η καλύτερη λύση για τον φορολογούμενο, όπως είπε η κυρία Νοβάκοφ. Εγώ θέλω να χρησιμοποιούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δημόσιο χρήμα. Διερωτώ με, είμαστε συνεπείς, μήπως μερικές φορές ζητούμε το αδύνατο, ε, να κάνουν τα αδύνατα δυνατά αυτές ε, οι υπηρεσίες, αυτοί οι οργανισμοί, ε, τους να θέτουμε νέα καθήκοντα χωρίς να τους δώσουμε νέους πόρους. Κάτι που αναφέρθηκε επίση Η συστηματική χρήση συμβασιούχων και η όλο και μεγαλύτερη χρήση εξωτερικών συμβούλων. Αυτό σημαίνει ότι οι θέση απασχόλησης ε, δεν έχουν μια σιγουριά. Δεν αφισβητώ την ποιότητά τους, έτσι, δεν αφισβητώ ότι κάνουν ποιοτική δουλειά, αλλά θα πρέπει να έχουν ένα χρονικό ορίζοντα πιο μεγάλο μπροστά του. Φυσικά αυτό που επιλέγετε είναι λιγότερο δαπανηρό. Αλλά θέλω να ρωτήσω όλους τους συναδέλφους για τη σκοπιμότητα αυτών των επιλογών μακροπρόθεσμα. Και τέλος, επειδή είμαι θα ήθελα να θέσω μία προκλητική ερώτηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τώρα που έχουμε κάποιο, κάποια εμπειρία και κάποιο χρόνο πίσω μας, χρησιμοποίησαμε ε, σωστά τους οργανισμούς. Μήπως υπάρχουν πολλοί οργανισμοί. Ρωτάω τον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου. Μήπως δεν υπάρχουν αρκετοί. Υλοποιούν την αποστολή τους. Μήπως θα έπρεπε να αναθέσουμε αυτές τις αποστολές σε εξωτερικούς φορείς, σε εξωτερικούς οργανισμούς. Είναι λίγο προκλητική ερώτηση, αλλά μετά την ανάγνωση της έκθεσής σας μου έρχεται αυτό το ερώτημα στο μυαλό. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Και στο τέλος να δώσω το λόγο στον κύριο Κούς και μετά έχουμε τον κύριο Λεζερή. Μέχρι τις 4 έχουμε την ώρα για να απαντήσουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Χολμάιερ. Πολύ σε αυτές οι εκθέσεις και πολύ ενδιαφέρουσες και οι ερωτήσεις και νομίζω ότι ε, πρέπει να είμαστε άτεκτοι για να έχουμε τι σωστέ απαντήσει στα σωστά ερωτήματα και καταρχά να απευθύνω ένα μεγάλο έπαινο καταρχάς γιατί έγινε πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά τι εκθέσει αυτέ. Και νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάποιο βασικό, κάποια βασική εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά την ποιότητα της εργασίας. Παραμένουν κάποια ερωτηματικά ωστόσο και όπως είπαν και οι συνάδελφοι ο κ. Μπολιέ έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Αναρωτιέμαι γιατί υπάρχουν λοιπόν τόσο πολλά, τόσο πολλοί οργανισμοί και δεν είναι μόνο και οργανισμοί. Έχουμε και τις ε, υπηρεσίες, ε, τις κοινέ εταιρείε και τα κοινές επιχειρήσεις. Οι συνέργειες που υπάρχουν αξιοποιούνται. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τα κοινά στοιχεία σε ό,τι αφορά τα κοινά προγράμματα, σε ό,τι αφορά τις κοινέ ε, εγκαταστάσεις ε, και τα κοινά προγράμματα πληροφορικής. Τι γίνεται με τα κτίρια, μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάποια κοινά κτίρια και το καθεξής. Και τι γίνεται με άλλα με άλλες εγκαταστάσεις, στην ΕΑΖΟ για παράδειγμα, όταν βρίσκεται κάπου στο εξωτερικό. Υπάρχουν και εκεί ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όπως για παράδειγμα η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αξιοποιούνται οι ευκαιρίες που υπάρχουν για να υπάρχουν κάποιες συνέργειες ή μήπω δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Δεν ξέρω κιόλα. Αλλά αυτό φαντάζομαι ότι θα εξοικονομούσε πολλά χρήματα και θα μπορούσαν πολλές ευκαιρίες να αξιοποιηθούν τον τρόπο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. λέει ο πρόεδρο. Έχουμε εδώ πέρα την ΕΑΖΟ. Να δώσω λοιπόν το λόγο καταρχάς στον κύριο Χάνσεν. Και στο τέλο ε, τον κύριο Λεζερή από την Frontex. Θα προσπαθήσω να ξεκινήσω με τις πιο γενικές ερωτήσεις. Ε, και πριν κλείσει αυτό το σημείο θα κάνουμε και μια καταληκτική παρατήρηση από πλευρά δικτύου οργανισμών. Λοιπόν, για, το, για τη γενική ερώτηση ότι μειώνεται ο προπολογισμό, αυξάνονται τα καθήκοντα, πώ θα το αντιμετωπίσουμε. Ένα από τα καθήκοντα που το δίκτυο των οργανισμών έχει είναι συνεχώς να ανταλλάσσει εμπειρίες για το πώς θα γίνουν πιο αποτελεσματικοί, για το πώς θα υπάρξουν συνέργειες, σε ποιους έξουν τρόπους εργασίας, και πώς θα πετύχουμε περισσότερα με λιγότερα χρήματα. Ε, γι' αυτό έχουμε το δίκτυο. Είναι πάντα στο μυαλό μας αυτό. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από το δικό μου οργανισμό, αλλά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Ε, όταν, ας πούμε, είναι κοντά οι οργανισμοί, ε, μπορούν να μοιραστούν, ας πούμε, τις συμβάσεις, τους διαγωνισμούς. Εμείς έχουμε κάποια αρμοδιότητα για κάποια είδη δεδομένων η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Τροφίμων ε, έχει σφιχτές προθεσμίες για, ένα νέο, για μια νέα νομοθεσία και τη βοηθάμε για να εφαρμόσει τη δική της νομοθεσία. Ε, και πώς το κάνουμε αυτό, γιατί γνωριζόμαστε μεταξύ μας, ξέρουμε τι δύναμη έχει ο καθένας και όταν έχουμε ευκαιρία να το κάνουμε, την αρπάζουμε. Δεν είναι ότι θέλουμε να κάνουμε περισσότερη δουλειά μόνο, είναι ότι θέλουμε να δώσουμε υπηρεσία στους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε και μια τελεία. Στις δύο τελευταίες συνεδρίασεις του δικτύου ε, συνειδητοποίησαμε ότι φτάνουμε αυτό το όριο. Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε αυτά που μας αναθέτουν, που είναι όλο και περισσότερο τα κάνουμε, χωρίς νέους πόρους. Ως δίκτυο πιστεύουμε ότι σχεδόν έχουμε φτάσει αυτό το όριο. Ίσως υπάρχουν κάποια περιθώρια για κάποιους οργανισμούς. Εμείς, ας πούμε, στον οργανισμό μας αυξήσαμε τον όγκο εργασίας, τα βασικά μας καθήκοντα, κατά 50% χωρίς επιπλέον πόρους. Αυτό το εξασφαλίσαμε μειώντας δραστηριότητες, κάνοντας, ε, βάζοντας προτεραιότητες, ε, δεν κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μας υποχρεώνει η νομοθεσία να τα κάνουμε. Ε, δεν πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε καινούργια πράγματα αν δεν μας δοθούν περισσότεροι πόροι και ξέρω ότι και άλλοι συνάδελφοι έχουν την ίδια άποψη. Επομένως, σας λέμε, ναι, μπορεί να έχουμε πρόβλημα αν συνέχεια υπάρχουν περικοπές και υπάρχουν και περισσότερες προσδοκίες. Φυσικά, εάν οι προσδοκίες προς εμάς μειωθούν, πολιτικό πώ μειωθούν, τότε δεν χρειαζόμαστε περισσότερου πόρου. Αλλά αν οι προσδοκίε για εξυπηρέτηση του πολίτη ε, είναι όλο και μεγαλύτερε, τότε θα πρέπει να μα δοθούν οι επιπλέον πόροι. Αυτό το λέω γενικά, έτσι. Θα πρέπει να δούμε τι λεπτομέρειε. Τώρα, για τι πιο συγκεκριμένε ερωτήσει. Κάποιε από τι πολιτικέ, σε ό,τι αφορά του ε, καταγγέλλοντε, την ε, παρα... παρενόχληση και τι οικονομικέ ατασταλίε, δεν μπορώ να μιλήσω εξ του δικτύου γιατί δεν ρωτάμε τους πάντες. Ξέρω ότι πολλοί οργανισμοί κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, ε, έθετα αυτό το ερώτημα στους συναδέλφους και οι περισσότεροι μου λέγανε ότι υπάρχουν τέτοιες πολιτικές ε, για αυτά τα θέματα. Ε, εμείς έχουμε, ας πούμε, θέμα πολιτικές για τη διοντολογία, για τους καταγγέλλοντες, τους whistleblowers και τα θέματα παρενόχλησης. Και όταν κάποιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά, μας, τα καθήκοντά του στην, στον οργανισμό μας, τον ε, περνάει από αρχικά μαθήματα για αυτά τα θέματα και κάθε τόσο περνάει από επαναληπτικά μαθήματα. Ως δίκτυο έχουμε συμβούλους για την παρενόχληση. Ε, είναι εμπιστευτικέ αυτές οι επαφές με το προσωπικό των συμβούλων. Εγώ έχω τακτικές συνεδριάσεις με αυτούς τους ε, συμβούλους και ενημερώνομαι για το ποια είναι τα προβλήματα και δουλεύουμε με τους ανθρώπους, ε, στους ανθρώπινους πόρους για να τα αντιμετωπίσουμε. Φυσικά υπάρχουν επίσημες διαδικασίες, τις χρησιμοποιούμε στον οργανισμό μου και αυτό δείχνει που παρότι δυστυχώς ε, ορισμένοι αισθάνονται ότι παρενοχλούνται, το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι διαδικασίες σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε. Γενικά κάνουμε αυτή τη δουλειά αλλά δεν μπορώ να εκπροσωπήσω εδώ πέρα όλου τους οργανισμούς. Τώρα, κάποιες άλλες ε, ερωτήσεις για το ΕΚΑ και την ε, εξωτερική ανάθεση. Τα βασικά μας καθήκοντα εμεί τα κάνουμε. Τις εξωτερικές αναθέσεις τις κάνουμε για θέματα πληροφορική. Είμαστε σε μια ψηφιακή εποχή. Έχουμε χιλιάδες εταιρείε οι οποίες ε, πρέπει να μιλήσουν μαζί μας, πρέπει να μας υποβάλουν πληροφορίες δεκάδες χιλιάδες, για δεκάδες χιλιάδες πράγματα. Επομένως, ε, η πληροφορική είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για μας. Ε, και υπάρχουν σύμβουλοι που έρχονται και ε, εξετάζουμε μήπως αναθέτουμε εξωτερικά τις, τα βασικά μας καθήκοντα. Αλλά ο σύμβουλος αυτός είπε ότι κάνουμε σωστές αναθέσεις. Δεν κάνουμε εξωτερική ανάθεση των βασικών καθηκόντων μας. Ε, και παρόλα αυτά είμαστε εντάξει και με θέματα πληροφορικής. Ε, για να για το θέμα το, του οικονομικού μας μοντέλου και κατά πόσο είναι βιώσιμο, ε, το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι ότι τα έσοδα από τα τέλη δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εκ των προτέρων με ακρίβεια. Είναι συν πλην 10 ε, εκατομμύρια ευρώ. Όταν το συνολικό προπολογισμό μα είναι 110 εκατομμύρια ευρώ, καταλαβαίνετε ότι το 10 εκατομμύρια είναι μεγάλο νούμερο ε, έχουμε πρόβλημα με την εκτίμηση των τελών και να, για να έχουμε μια σταθερή χρηματοδότηση. Είναι κάτι που το εξετάζουμε πολύ στενά με τους συναδέλφους από την Κομισιόν. Φυσικά εξαρτάται από την Κομισιόν για να γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά εμείς έχουμε ιδέες. Είτε να αλλάξουμε το μοντέλο των, της χρηματοδότησης μέσω τελών, να χρηματοδοτούμαστε, ε, να χρηματοδοτούμαστε ναι μεν από τα τέλη, αλλά τα τέλη να πηγαίνουν κατευθείαν να εισπράττονται από την Κομισιόν. Θα πρέπει να γίνουν αυτές οι συζητήσεις. Έχουν, γίνει, έχουν ξεκινήσει. Μέχρι στιγμής ήταν πολύ καρποφόρες με τους συναδέλφους της Κομισιόν. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που αφορούσαν το ΕΚΑ. Ο Λεζερή, ο κ. Λεζερή ε, θα μου απαντήσει. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ο κύριος Λεζερή από τη Frontex θα απαντήσει τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιβεβαιώνω ότι στη Frontex έχουμε πολιτική για τους καταγγέλλοντες και έχουμε και τη σεμινάρια κατάρτιση για το προσωπικό όταν αναλαμβάνει καθηκοντά του κανείς στην Frontex. Έχουμε πολιτικές κατά της παρενόχλησης και μόλις έχουμε διορίσει ε, συμβούλους εμπιστευτικότητας ε, και αυτοί λαμβάνουν μάλιστα κατάρτιση από μια αρμόδια εταιρεία, εξωτερική εταιρεία. Τώρα, για το ότι εξαρτώμαστε από συμβασιούχους. Αυτό είναι κοινό σε, πολλές, ε, σε πολλούς οργανισμούς, ειδικά όταν ε, κυριαρχούνται από θέματα πληροφορικής. Υπάρχει ένα βασικό θεμελιακό ερώτημα ε, για θέματα πληροφορικής. Όταν μιλάμε για τις πολιτικές εσωτερικών, όπου έχουμε τεράστια συστήματα πληροφορικής, είναι λογικό ότι ο οργανισμός εταίρος μας είναι η Ιουλίσα. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη όμως μικρότερων δικτύων πληροφορικής, τότε εκεί πρέπει να απευθυνθούμε σε εξωτερικές εταιρείε, να κάνουμε εξωτερική ανάθεση. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Ε, αν κάνουμε προσλήψεις, αν θέλω να προσλάβω, ας πούμε, στη Βαρσοβία με το συντελεστή διόρθωση που είναι 68 αυτή τη στιγμή, αν θέλω να προσλάβω πληροφορικάριους υψηλού επίπεδου, θα δυσκολευτώ. Γιατί οι περισσότεροι θέλουν να πάνε στην ιδιωτική αγορά, να βρουν μια δουλειά σε ένα κράτος μέλος όπου έχει υψηλούς μισθούς. Σε ό,τι αφορά το αμύφα για τη Frontex. Το Ταμείο ε, Ασύλου και Μετανάστευσης και το Frontex, το ΑΜΙΦ δηλαδή, το ΑΜΙΦ ε, αποφασίστηκε πριν ενισχυθεί η εντολή της Frontex. Αυτό που κάναμε με τη Γενική Διεύθυνση Home της ε, χρηματοδότησης της Κομισιόν είναι να μην υπάρχει κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης. Και επίσης συντονίζουμε την προσέγγιση μας η Frontex μαζί με το ΑΜΙΦ. Αλλά εμείς ως οργανισμός ασχολούμαστε με δράσεις επιστροφής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάνουμε και ε, επιχειρησιακή στήριξη. Σε ό,τι αφορά, δίνουμε επιχειρησιακή ε, στήριξη. Σε ό,τι αφορά κάποια επεισόδια που παρατηρήθηκαν κάτι διάφορα επιχειρήσεων επιστροφών. Επιστρέψαμε το 2018 πάνω από 1.400, ε, συγγνώμη, πάνω από 14.000 άτομα. Αν τα ε, συγκρίνετε με, τις, ε, με τα επεισόδια που είχαν τα κράτη-μέλη, μια χαρά είμαστε. Μόνο τρεις, ε, σε τρία επεισόδια κάποιοι συνοδοί τραυματίστηκαν. Δεν είναι ψηλό το νούμερο. Φυσικά πάντα μπορούμε να βελτιώσουμε τις διαδικασίες, αλλά δεδομένου ότι είναι πολύ περίπλοκες οι διαδικασίες, μερικές φορές έχουμε συνοδούς διαφορετικών εθνικοτήτων. Μερικές φορές υπάρχουν προβλήματα γλωσσικά. Και το νομικό καθεστώ επίση είναι περίπλοκο. Το να έχουμε τρία επεισόδια δεν είναι τίποτα μόνο στι ε, περιπτώσει αυτέ επιστροφών. Για τον τεχνικό εξοπλισμό. Θέμα που έθεσε ο εισηγητή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα σκάφος από τη Λετωνία Είχαμε ένα σκάφο από τη Λετωνία. Αυτό το θέμα το συζήτησε και το ελεγκτικό συνέδριο. Το συνοδευτικό έγγραφο που υποβλήθηκε από το κράτος μέλος, ισχυριζόμενο, ε, ζητώντας την, ε, τα έξοδα, το έγγραφο αυτό έλεγε ποιο είναι το συνολικό κόστος, έλεγε ποια είναι η περίοδος που χρησιμοποιήθηκε, ε, τα ποσά που, χρειάζονται, εννέα βάρδιες και άλλα ποσά και, άλλες, και άλλα έξοδα. Έχουμε ένα σαφή κατάλογο με, όλο, με όλα τα επιμέρους κόστη. Και αυτό το υπέγραψε ο, ο διοικητής της ε, λετονικής ε, συνοριοφυλακής. Νομίζουμε ότι επαρκεί αυτό. Για να σας εξηγήσει ποιο είναι το κόστος και να μας δώσει και την διασφάλιση ότι ήταν αρκετά τεκμηριωμένη η αίτηση αυτή για επιστροφή εξόδων. Ε, για τη νέα πολιτική, για, τα ευαίσθη, για τις ευαίσθητες θέσεις, το, το εξετάζουμε αυτό το θέμα. Η δυσκολία είναι ότι ο οργανισμός μας αναπτύσσεται, μεγαλώνει, αλλάζει και άλλαξε πολύ τους τελευταίους 12 με 18 μήνες ε, και με την δημιουργία του νέου Ευρωπαϊκού Μόνιμου Σώματος θα έχουμε και νέες ε, ευαίσθητες θέσεις ή επιπλέον ευαίσθητες θέσεις σε ό,τι αφορά τις συνέργειες και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις κοινέ υπηρεσίες ή κοινά κτίρια με άλλους οργανισμούς. Ε, Παραδείγματο χάρη έχουμε ο αξιωματικούς συνδέσμους σε τρίτες χώρες όλοι βρίσκονται στα κτίρια, στα γραφεία των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, γιατί αυτοί οι αξιωματικοί βρίσκονται σε ένα γραφείο που τους τα δίνει δωρεάν το Υπουργείο Εσωτερικών του εν λόγω κρατούς μέλους. Ευχαριστώ τον κύριο Λεζερή. Παρακαλώ σεβασμό του χρόνου, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η κυρία Δεγκρεγκόρη έχει δύο λεφτά μόνο για να απαντήσει συνοπτικά στις ερωτήσεις. thank you very much Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα πρώτα σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και για τη θετική σας στάση, αξιότιμη κυρία Βουλευτέ. Είναι μεγάλη μας τιμή να διαπιστώνετε κι εσείς ότι προσπαθούμε να βελτιωθούμε θα είμαι σύντομη, απαντώντας μία-μία τις ερωτήσεις. Ο κύριος Νοβακόφ έθιξε το ζήτημα των εθνικών εμπειρογνωμόνων. Μειώνονται. Μόνο 13% καλύπτουν τις κινήσεις μας. Δεν είναι καλό αυτό. Γιατί εμεί βοηθούμε περισσότερο τα κρατη Άρα, πρόβλημα. Αναντιστοιχεία και σύμφωνα με το πρόγραμμά μας συνέχεια ασχολούμεθα με τις αποβιβάσεις των μεταναστών έχουμε εννέα δράσεις ενώ έχουμε 1900 διασώσει και τα κράτη-μέλη μας βοηθούν όσον αφορά το προσωπικό τώρα αφορά τον έλεγχο για τις επιδόσεις μας, για ΕΚΑ και ΕΑΣΟ και τον συντονισμό. Για τον προϋπολογισμό τα είπε ο κύριος Λετζέρη. Ξέρουμε τι γίνεται με την κρηματοδότηση των κρατών μελών προς την ΑΜΙΦ. Και όταν εμείς κάνουμε επιχειρησιακά προγράμματα, και πρέπει να γίνει κάποια αξιολόγηση. Αυτό γίνεται πάντοτε σε συνεργασία με τα κρατημέλη, τα εμπλεκόμενα και σε συντονισμό με την Κομισιόν. Προσέχουμε να μην έχουμε ε, ε, επικαλύψεις. Αυτά και για τον προπολογισμό της ΙΑΖΟ τώρα όσον αφορά τα πυρσιακά μας δεδομένα στην Ελλάδα, τα στοιχεία και τα δύνατα σημεία εμείς έχουμε τα δικά μας στοιχεία και έχουν γίνει και αξιολογήσεις από τις υπηρεσίες. Και υπάρχει διαδικασία για τα σύνορα, επισημαίνονται τα δυνατά σημεία, άλλαξε τον Αύγουστο τη διαδικασία, γιατί άλλαξαν τη διαδικασία οι ελληνικές αρχές και έχουμε τώρα νέα νομοθεσία. Άρα έτσι θα πάει τώρα. Ρωτήσατε επίσης Καθώς να πρέπει να προσαρμοστούμε στις τρέχουσες ανάγκες και τι να σας πω, είπατε για την εντολή μας, το 10 πήραμε την εντολή μας και είναι παλιά. Δεν νομίζω ότι είναι έντολη που αντιστοιχεί στα σημερινά και στις ανάγκες των κρατών μελών. Γνωρίζω ότι έκλεισαν οι συνομοθέτες συμβιβασμό το 17 σε σχέση και με την ε, υπηρεσία εξωτερική δράση. Μετά είχαμε τον μπλοκάρισμα με την νομοθεσία για το άσυλο, αλλά με μια νέα συμφωνία η Κομισιόν ίσως προτείνει επαναξιολόγηση της εντολής. Και νέο κανονισμό. Οπότε ελπίζουμε ότι θα αναβαθμιστούμε. Πάντως, όσον αφορά την εποπτεία. Θα πρέπει τουλάχιστον να επιτρέπει εντολή να αξιολογούμε τους κινδύνους και να κάνουμε προγνωστικά με κάποιο σύστημα έγκαιρης προδοπής προς τα κρατη σε σχέση με το άσυλο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γρηγόρη και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, μας το Ελληνικό Συνέδριο, αλλά έχει καταφτάσει ο επίτροπο, Θα τον καλωσορίζω. Αν θέλετε, κύριε Σάντσο, έχετε δύο λεπτάκια να πάρετε το λόγο και στο τέλο και ο συγκεκριτή μα και μετά να περάσουμε κατευθείαν στο επόμενο θέμα τη ημερήσια διαταξή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μια και άκουσα κάποιε ερωτήσει από τον κύριο Μπογέ. Ε, κοιτάξτε, εμένα μου αρέσουν αυτέ οι προκλητικέ ερωτήσει, αλλά να απαντήσω στα σοβαρά σας ε, επιστώ την προσοχή σας στον αριθμό και τη γεωγραφική κατανομή των οργανισμών. Σελίδα 8 της σύνοψης της έκθεσής μας. Κοιτώντας το χάρτη αυτό, η πρώτη εντύπωση που μου δίνεται είναι ένας ε, χάρτης ο οποίος έχει πολλές ε, πινέζες στον τοίχο. αυτές οι Πινέζες κρατούν μαζί την Ένωση, ενωμένη. Και κατά δεύτερον, να συμφωνήσω με τον κύριο Νόβακοφ, το οικοσύστημα αυτό των οργανισμών, 40 και πλέον στον αριθμό, παίζει πολύ πιο σημαντικό ρόλο. Όχι μόνο για να συγκρατήσει την ε, ενότητα της Ένωσης, με τόσο μικρό αριθμό ανθρώπων και τόσους λίγους πόρους. Είναι πραγματικά μαγικό. Που μπορούμε να το πετύχουμε μόνο μαζί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πάλι τους οργανισμούς, ευχαριστώ και τα μέλη της Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δίνετε τόση σημασία στα σημαντικά αυτά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να ακούσουμε τον κύριο Μπρουντζίτσκι, τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και όντως, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την πολύ χρήσιμη αυτή ανταλλαγή απόψεων και τις ερωτήσεις αυτές που νομίζω ότι κάλυψαν πολλά από τα κοινά που είχαμε στο επόμενο θέμα της... Ε, θα τα ξαναπούμε μάλλον στις ε, 21 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Θα είναι η επόμενη ευκαιρία που θα έχουμε να αλλάξουμε απόψει. Και στις 29 είναι η προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών. Και μετά θα έχουμε και φυσικά την συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Νίκη Πρόεδρος. Ολοκλήρωμε, λοιπόν, ε, ευχαριστήσω, λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους τους ε, επικεφαλής και εκπροσώπους των οργανισμών. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και να περάσουμε στο επόμενο θέμα, στην ημερήσια διάταξη. Απαλλαγή 2018, Γενικός προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι λοιπόν που καλώς ορίζω και πάλι τον ε, Επιτροπό τον κύριο Σμίτ, ο οποίος έχει το χαρτοφυλάκιο για τις θέσει απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα στην νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συνεχίσω να μιλώ μέχρι ότου εξέλθουν από την αίθουσα αυτοί που είχαν έρθει για το προηγούμενο σημείο για να μην σας ε, ενοχλήσει ο θόρυβος. Ich freue mich, dass in diesem Zusammenhang äh, das mit... Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε μαζί μα και μέλη του ηλεκτρικού συνεδρίου, τον κύριο Μέρφυ και την ομάδα του. Καλώ ορίσατε κι εσεί. Θα έχουμε 90 λεπτά στη διάθεσή μα να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Να ακούσουμε τον Επίτροπο την ελεκτικό συνέδριο και μετά θα μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς ερωτήσεις ως βουλευτές. Να δώσουμε καταρχάς ε, τον εκπρόσωπο του ελεκτικού συνεδρίου, τον κύριο Μέρφυ, για να μας παρουσιάσει την έκθεση του και μετά να ακούσουμε και τον Επίτροπο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε και κύριοι Επίτροπε. Sorry. No, Sorry, ladies. Listen. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη, ε, με μεγάλη χώρα έρχομαι εδώ στην Επιτροπή για να παρουσιάσω το κεφάλαιο 6 της ε, ετήσιας έκθεσης του 18. Ε, συναντώ τον Επιτρόπο Σμιτ για πρώτη φορά του εύχομαι καλή επιτυχία για το πολύ σημαντικό αυτό κομμάτι πολιτικής της Κομισιόν. Ε, το κεφάλαιο αυτό είναι η ειδική αξιολόγηση για τις δαπάνες οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής υπό το πουδουπού υπότιτλος 1β και καλύπτει ε, και τα κονδύλια που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης ε, και, δηλαδή απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις και η Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο δεν κάνει χωριστή αξιολόγηση για, τα, ε, για το κοινωνικό ταμείο και την πρωτοβουλία απασχόληση των νέων. Ε, δεν το έχει κάνει από, το, από την ετήσια έκθεση του 2014. Επομένω, είναι αναπόφευκτο ότι θα υπάρξουν επικαλύψει ανάμεσα στην παρουσίασή μου σήμερα και σε αυτή που έγινε στι 11 Νοεμβρίου ε, στην ακρόαση για την περιφερειακή πολιτική. Ο στόχο είναι διτό να συνεισφέρουμε στην ε, συνολική διασφάλιση, ποιότητα, ε, διασφάλιση ε, ποιότητας και να αξιολογήσουμε το νέο έλεγχο και το νέο πλαίσιο διασφάλισης για την περίοδο 14-20. Αυτό το νέο πλαίσιο δίνει στα, στις αρχές των κρατών μελών, ή μάλλον το λάθος μάλλον είναι κάτω από 2%. Η Κομισιόν δέχεται ότι οι δαπάνες ε, είναι σωστές και ο στόχος είναι <clears throat> να αυξάνουμε την τακτικότητα τις τακτικές πληροφορίες υπό το νέο αυτό πλαίσιο ελέγχου και διασφάλισης και να μειώσουμε το διοικητικό άχθος. Για φέτος ε, εξετάσαμε 220 συναλλαγές, εκ των οποίων 69, περίπου το 1 τρίτον, αφορούσαν τη Γενική Διευθύνση Απασχόλησης. Ε, μιλάμε για συναλλαγές που τα κράτη-μέλη είχαν ελέγξει προηγουμένως και κάναμε μία αναθεώρηση του καταλόγου και των ελέγχων που κάνουν για να ε, επιβεβαιώσουμε τις απόψεις τους. Ε, είχαμε 36 λάθη, 18 αφορούσαν το, ε, το Κοινωνικό Ταμείο και την Πρωτοβουλία Απασχολήσεων των Νέων και που δεν είχαν εντοπίσει οι αρχές. Λαμβάνοντας υπόψη τα, τα 60 λάθη που είχαν εντοπίσει πριν οι αρχές, καθώς και τις διορθώσεις των κρατών μελών για 340 εκατομμύρια ευρώ, εκτιμούμε ότι το ποσοστό σφάλματος για το 1β του πουδουπού είναι μικρότερο από πέρυσι. Το 2017 ήταν περίεργη χρονιά. Μόνο 17 ε, κράτη-μέλη είχαν υποβάλει ένα χαμηλό βαθμό δαπανών και το ποσοστό σφάλματος ήταν υψηλότερο από τη συνήθως φέτος. Ε, οι λάθος ε, δαπάνες και η παραβίαση των κανόνων που αφορούν συνήθως ε, το ERDF ε, και αφορούσαν κυρίως τα λάθη. Τονίσαμε ότι οι εθνικοί κανόνες είναι περίπλοκοι και θα πρέπει να απλουστεύσουμε λίγο τα μέτρα. <laughs> Ο δεύτερος στόχος της, ε, του ελέγχου του 18 ήταν να αξιολογήσουμε το νέο πλαίσιο ε, διασφάλισης και ελέγχου 14-20 και να καλύψουμε τις δραστηριότητε των κρατών μελών και της Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο στόχο, που ήταν η αξιολόγηση της δουλειάς των κρατών μελών και των αρχών τους, φέτος αξιολογήσαμε 15 από, 100, τις 126 ελεγκτικές αρχές και βρίσκουμε ότι οι ελεγκτικές αρχές εξέδωσαν ε, καθαρές νομοδοτήσεις για τις παρατυπίες, δηλαδή πιστοποιούν ένα μικρό ε, σφάλμα κάτω του 2%, ενώ εμείς βρήκαμε ότι ήμασταν πάνω από αυτό το κατόφλι του 2%. Ε, αυτό συνέβη για 8 ε, α, από τις 8 από τις διασφαλίσεις ποιότητα. Η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης έχει αντίστοιχα προβλήματα στην ε, τήση έκθεση δραστηριοτήτων, όπου 30% 11 από τα 36 προγράμματα των OP που θεωρούν ότι είναι υποκίνδυνο και ελέγχθηκαν, ε, έχουν αναφερθεί λάθος, ε, με λανθασμένο ποσοστό σφάλματος και ήταν πάνω από το 2%. Επίσης βρήκαμε διάφορες αδυναμίες ό,τι αφορά τη δουλειά που έκαναν οι ελεγκτικές αρχές. Ε, αυτές αφορούν την ε, δειγματοληψία και παρά τις ε, βελτιώσεις υπάρχουν προβλήματα με το πεδίο εφαρμογή, την ποιότητα και την τεκμηρίωση της δουλειάς τους. Γι' αυτό έπρεπε να, ξανακάνουμε 64, να ξαναδούμε 64 συναλλαγές σε σχέση με 121 πέρυσι που είχαμε ξαναδεί, μεταξύ των οποίων 48 σε επιτόπιες επισκέψεις κάναμε σε δικαιούχου, ενώ πέρυσι είχαμε κάνει 80. Αυτό δείχνει μια συνολική βελτίωση. παρόλα αυτά, απαιτεί επιπλέον πόρου και οδήγησε σε πλέον άχθο για κάποιου ε, δικαιούχου. Α δούμε τώρα την αξιολόγηση τη δουλειά που έκανε η Κομισιόν. Τα αποτελέσματα τη δουλειά τη Κομισιόν είναι η βάση για να καθορίσουμε το ποσοστά σφάλματο και τις ε, επιφυλάξεις στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Ε, Ξετάσαμε το ποσοστό σφάλματος για την οικονομική χρονιά 2016-2017, όπου τα έξοδα ήδη είχαν ελεγχθεί με βάση το νέο κύκλο ελέγχου. Ε, το χειρότερο σφάλμα του 2,3% δεν ήταν οριστικό όταν η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης ε, δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για τα πεπραγμένα της τον Ιούνιο του 2019 πιθανές διορθωτικές δράσεις για 47 από τις 141 ούπης ε, συνεχίζονται ακόμα και αυτό το ποσοστό σφάλματος είναι μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό λόγω της μεθοδολογίας της Κομισιόν. Ένα άλλο σημαντικό ποσοστό σφάλματος για τη Γενική Διεύθυνση Επασχόλησης είναι ο κίνδυνος κατά την πληρωμή που, που παρακολουθεί την αρχή του δημοσιονομικού κανονισμού και συνδέεται με τις δαπάνε για το κοινωνικό ταμείο και την πρωτοβουλία απασχόληση των νέων του 18. Αυτές οι δαπάνε δεν έχουν ε, υποβληθεί στο νέο κύκλο ελέγχου όταν δημοσιεύτηκε η ετήσια έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης και ο κίνδυνο ε, κατά την πληρωμή του 2,1% είναι εκτίμηση και μπορεί να υποστεί διορθώσει και να θα επαληθευτεί βέβαια. Κυρίε και κύριοι, Δεδομένων των ε, λήψεων στο νέο πλαίσιο ελέγχου και διασφάλισης που σας ανέφερα, δεν μπορούμε να βασιστούμε στη δουλειά που κάνουν τα κράτη-μέλη και οι ελεγκτικές τους αρχές αυτή τη στιγμή ή τα ποσοστά ασφάλματος που παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης. Κάναμε τρεις συστάσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση στο μέλλον. Η Κομισιόν τις δέχτηκε και επίσης παραπέμπουμε στις συστάσεις που κάναμε πέρυσι και που αφορά θέματα τα οποία και προβλήματα που ξαναβρήκαμε και φέτος. Αγαπητοί βουλευτέ, είναι κρίσιμο να ξοδεύουμε τα κονδύλια τη Ένωση με βάση του κανόνε. Είναι ζωτική σημασία, λόγω του ότι έχουμε πολύ λίγου δημοσιονομικού πόρου, να έχουμε θετική επίπτωση, υλοποιώντα δηλαδή του στόχου και να πετυχαίνουμε αποτελέσματα με τα λεφτά που ξοδεύουμε. Αξιολογήσαμε σε χωριστό τμήμα του κεφαλαίου 6 στοιχεία των επιδόσεων των κρατών μελών βρήκαμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν μηχανισμούς ε, παρακολούθησης για να καταγράφουν ε, τι πληροφορίες για τις επιδόσεις, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οι αρχές δεν έχουν τέτοια αποτελέσματα ε, δικτών σε επίπεδο έργου και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχουμε καν τέτοιους δείκτες. Επίσης, κάποια project, κάποια έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί δεν έχουν πάντα υλοποιήσει τους στόχους τους. Ελπίζω ότι αυτά τα απορίσματα και τα συμπεράσματα να είναι χρήσιμα για την Επιτροπή σας και για την ε, Κομισιόν. Ε, η σημασία αυτής της πολιτικής απεικονίζεται ε, από το γεγονός ότι 13 ειδικέ εκθέσεις και 6 ανθεωρίες που αφορούν θέματα συνοχής δημοσιεύθηκαν από το Ελεκτικό Συνέδριο το 2018 και το 19 μέχρι σήμερα. Θα ήθελα να τελειώσω την παρουσίασή μου τονίζοντας ακόμα μια φορά ότι τα σφάλματα που εντοπίζουμε οφείλονται και οφείλονται στην μη συμμόρφωση με τους τρέχοντες κανόνες και δεν σημαίνει κατά ανάγκη ε, σπατάλη πόρων, γιατί αυτά τα έργα τρέχουν ακόμα και μπορεί όταν τελειώσουν να έχουν ε, επιτύχει θετική επίπτωση και να έχουν ε, υλοποιήσει τους στόχους τους. Ευχαριστώ την ε, εισηγήτρια την κυρία Χολμάιερ για τις ανταλλαγές απόψεων και την Κομισιόν για την επικοδομητική σχέση εργασίας που είχαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι πάντα εύκολη, γιατί είναι πολύ περίπλοκος αυτός ο τομέας πολιτικής και μερικέ φορέ κάνουμε και επαγγελματικέ αξιολογήσει και κρίσεις. Τέλος, να πω και κάτι προσωπικό. Αυτό το κεφάλαιο Ε, για αυτό το κεφάλαιο μας ε, βοήθησε ένας ε, λιγκτής ο οποίος ε, ήταν καταπληκτικός και δυστυχώς πέθανε ευνίδια πριν από τρία, τρεις εβδομάδες. Τώρα θα ήθελα να ακούσω την παρουσίαση του Επιτρόπου Σμιτ και τις ερωτήσεις των βουλευτών. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή συνεργασία και για τις πολλές ε, πληροφορίες, ε, για τις πολλές πολλές ερωτήσεις που κάναμε και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουμε να θέτουμε τέτοιες ερωτήσεις ε. Πρόκειται για μια διαδικασία αντίχω τέλο ε, σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και των εισηγητών. Θα σα καλωσορίσω λοιπόν και πάλι, κύριε Επιτροπέ, και θα σα δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε. Καταρχά, να σα ευχαριστήσω για την ε, εισαγωγή σας και για την ε, η υποδοχή σας αξιότιμοι βουλευτές, αξιότιμο ελεκτικό συνέδριο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια που μας ε, είπατε. Είναι τιμή μου που παρουσιάζομαι εδώ λοιπόν στην Επιτροπή και ε, τη δική σας όπως και στις άλλες επιτροπές ε, για να παρουσιάσω τα στοιχεία αυτά τα οποία αφορούν τα τελευταία χρόνια και τα όσα έγιναν. Να μιλήσω καταρχάς για τα όσα έκανε η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναλαμβάνω λοιπόν τα καθήκοντα εδώ πέρα και να σας μιλήσω και για το δικό μου πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στο, στην επιστολή αποστολή και στις γενικές κατευθυντηρίες γραμμές τις οποίες εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πρότεινε ένα συνεκτικό πλαίσιο για την κοινωνική πολιτική και σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό των εξόδων και των δαπάνων για τα επόμενα έτη. Και σύμφωνα με όσα δηλώθηκαν στον Κατεμπορό το 2017, προκειμένου η κοινωνική Ευρώπη να παραμείνει προτεραιότητα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να, να δημιουργήσουμε μία Ευρωπαϊκή Ένωση και μία κοινωνική οικονομία πιο ανταγωνιστική, πιο δίκαιη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει σύγκληση οικονομική αλλά και κοινωνική Μία λοιπόν από τις ε, αποστολές της Επιτροπής αυτής θα είναι τα υλοποίηση όλα αυτά. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, παρουσίασε μια λοιπον απο τις αποστολες της επιτροπης αυτη θα ειναι τα υλοποιήσει πρωτοβουλειών ε, που θα ενισχύσουν την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα έτη. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν συγκεκριμένα μία νομοθετική πρόταση προκειμένου κάθε εργαζόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει ένα ίσο και δίκαιο μισθών, μια προστασία από την ανεργία και μια ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, όπως ε, η εγγύηση για, τα, για τους νέους αποδέχτηκε πολύ αποτελεσματική στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας. Θα συνεχίσουμε να την προωθούμε και θα την προσαρμόσουμε. Θα ενημερωθεί επίσης η στρατηγική για τις δεξιότητες και τα προσόντα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη μετάβαση την κλιματική αλλά και την τεχνολογική. Επίσης σημαντικό είναι η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή για την Εργασία να τεθεί ε, σε λειτουργία και να στηθεί στα πόδια της σύντομα και γρήγορα. Θα συνεχίσω να τονίζω τα βασικά οικονομικά εργαλεία τα οποία έχω στη διάθεσή μου, το Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το EFS λοιπόν ε, χρησιμοποιήθηκε και αξιοποιήθηκε με πολύ ικανοποιητικό τρόπο από την προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρξουν επενδύσεις ε, στους εργαζομένους και να δοθεί βοήθεια στους ε, ανέργους και κυρίως του μακροπρόθεσμα ανέργους. Ε, το EFS λοιπόν ε, έδωσε 14 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν από το 2014 240.000 άτομα εργαζόνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραπάνω και πρόκειται για το πιο χαμηλό επίπεδο ανεργία εδώ και πολλά χρόνια, από το 2000 και μετά και προσπαθούμε να μειώσουμε περαιτέρω αυτό το ποσοστό. Έχει λοιπόν βοηθήσει το ESF 26 εκατομμύρια ανθρώπους και μακροπρόθερμα αργών. Περίπου 6 εκατομμύρια, 2,6 συμμετέχοντες και 1,4 ήταν σε ε, διαδικασίες και ενεργείες εκπαίδευσης. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων που αποτελεί το βασικό μας εργαλείο για την χρηματοδότηση και τη βοήθεια προς τους νέους για να έχουν πρόσβαση στις απασχόληση και στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση έχει υποστηρίξει 2,7 εκατομμυρία νέους μέχρι τη τέλη του 2018. Οι υπηρεσίες λοιπόν αυτές δίδονται ε, μονίμως για να εξασφαλίσουν ότι κάθε ευρώ το οποίο δαπανάτε έχει αποτέλεσμα. Έχουμε διαπιστώσει λοιπόν μια σημαντική βελτίωση τη ε, νομιμότητα και τη κανονικότητα των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την περίοδο της ε, προγραμματισμού 2007 με 2013 το ποσοστό σφάλμα το οποίο ήταν σε δεκαδικα διπλά ήταν πλέον μεταξύ 3 έως 5% μιας και πρόκειται Πρόκειται για ένα υψηλό ποσοστό σφάλματος, αλλά σημαίνει ότι έχουν σημειωθεί σημαντική πρόοδο σε σχέση με του προκατόχου μου, στον λοιπόν το ίδιο. Και προφανώ αυτό αφήνεται και στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή σα, του ιδιαίτερου. Δύο είναι οι βασικοί οι λόγοι που εξηγούν αυτή τη βελτίωση. Καταρχά, έχει ε, απλοποιηθεί και διευκρινιστεί η νομοθεσία και τα συστήματα ελέγχου και υποπτίας έχουν ενισχυθεί. Αυτό μας δίνει ακόμα πιο μεγάλη σιγουριά για την πολιτική συνοχή και στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 έγιναν βασικές διευθετήσεις που μας επιτρέπουν να εξασφαλίζουμε καλύτερα τις δαπάνες μας. 20, 10% λοιπόν της ε, 100% για πολιτική αυστηρή, για την πολιτική τέτοιες αναστολών και για τη δυνατότητα να γίνουν ε, διορθώσεις οικονομικές μιας και τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου εντοπίζουν τέτοια σφάλματα. Κατά δεύτερον, στους ε, ελέγχους που έγιναν για την προερίοδο 2014-2020, για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εισαγάγει διατάξεις ε, για το αγλοποιημένο υπολογισμό του κόστους. Είναι λοιπόν ένα καινοτόμο σύστημα για να υπολογίζονται οι δαπάνε. και αυτό επιτρέπει να γίνεται πιο εύκολα και γρήγορα η επαλήθευση των οικονομικών διατάξεων σε ό,τι αφορά την οικονομική στρατηγική και μειώνει τον κίνδυνο ποσοτικοποιημένων σφαλμάτων όπως ε, επιβεβαίωσε τελευταία, τα τελευταία χρόνια το ελεκτικό συνέδριο. Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέδειξε ότι αυτό το κόστος καλύπτει περίπου το 30% του ΙΕΦΕΣ και αυτό δαπανάται από το 80% των προγραμμάτων του ΙΕΦΕΣ. Είμαστε πεπισμένοι ότι ο στόχος του 50% των συναλλαγών σε ό,τι αφορά το απροποιημένο αυτό κόστος θα επιτευχθεί στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο το οποίο με τη σειρά του θα σημαίνει ακόμα πιο σημαντική μείωση του ποσοστού σφάλματος. Όλες αυτές οι εργασίες λοιπόν που αποτυπώνονται στο ποσοστό σφάλματος ε, φαίνονται από τη μία προγραμματική περίοδο προς την άλλη. Ωστόσο, όπως προσέξατε πέρσι, για τις ε, πληρωμές του 2018 το ποσοστό σφάλματος έχει πάει από το 3% στο 5%. Όπως μας υπενθύμησε και το ελεκτικό συνέδριο. Γιατί λοιπόν αυξήθηκε έτσι από ό,τι φαίνεται, σε ό,τι αφορά τι πληρωμέ του 2018. Καταρχά, ο όγκο των δαπανών που ελέγχθηκε από το ελεκτικό συνέδριο ήταν πολύ πιο υψηλό από ό,τι το προηγούμενο έτη. 23,6 δις ευρώ ε, δαπάνες ελέγχθηκαν σε σχέση με 8 του 2017 δις σε ό,τι αφορά και το EFS και αυτό σημαίνει ότι το 2018 τα, οι δαπάνες ε, αυτές ε, ε, Μα προσθέθηκαν λοιπόν στις δαπάνες αυτές ε, σημαντικές πηγές σφαλμάτων. Το Εθνικό Συνέδριο σε διάφορες περιπτώσεις έχει ερμηνεύσει με διαφορετικό τρόπο την νομοθεσία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό υπογραμμίζεται στο πλαίσιο του επόμενου πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και είναι σαφές ότι οι κανόνες θα πρέπει να είναι όσο πιο ε, απλή γίνεται. Οι κανόνες λοιπόν που είναι πιο απλοί συνεπάγονται λιγότερο ποσοστό σφάλματος. Και επίσης να πω ότι το ποσοστό του σφάλματος δεν σημαίνει αυτόματα απάτη. Αυτό το διευκρινίζουμε, το είπε και το ελεκτικό συνέδριο προηγουμένω. Πρόκειται για ποσά τα οποία δαπανώνται, τα οποία δαπανήθηκαν μάλλον με τρόπο που δεν συνάδει απόλυτα με τι διατάξει, τι νομοθεσίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο εθνικό επίπεδο. Κυρίε και κύριοι, ακολουθούμε με σωστό τρόπο τι υποχρεώσει μα. Έχουμε αποτελεσματικότητα. Και αυτό για τους Ευρωπαίους πολίτες αποτελεί πραγματική υπεραξία. Το EFS Plus τώρα προστατεύει τις δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια τα επόμενα χρόνια. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να επενδύουμε πόρους και στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στις δεξιότητες και υπολογίζουμε στην υποστήριξή σας για να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και ξέρω ότι η υποστήριξή σας και η υποστήριξή του, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι το δεδομένο. Προσβλέπω λοιπόν σε συνεργασία μαζί σας τα επόμενα χρόνια για να υπάρχει μια Ευρώπη κοινωνική προς ε, όφελος και στην υπηρεσία του κάθε πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστούμε, κύριε Επίτροπε. Και για την αναδρομική παρουσίαση και για την παρουσίαση του τι θα γίνει στο μέλλον. Και τα δύο μας τα αναφέρατε. Ως εισηγήτρια, να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση. Μία πρώτη ερώτηση για τις χρηματικές, ε, για τις ε, διορθώσεις. Τι πόσο των ε, πόσων που ζητήθηκαν πίσω καταβλήθηκε πραγματικά. Δεν έχει απαντηθεί αυτό. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε αυτή την προφορική ερώτηση. Τι ποσό των 2,75 εκατομμυρίων επιστράφηκε. Αν δεν μπορείτε να απαντήσετε τώρα, μπορείτε να μας τα απαντήσετε και γραπτός. Αν δεν έχετε τα στοιχεία αυτά στην διάθεσή σας. Επίσης, τα κράτη-μέλη αποδέχτηκαν αυτές τις διορθώσεις και τα ποσά των διορθώσεων ή μήπως προσπαθούν να προσάγουν τις υποθέσεις στο δικαστήριο. Έχουν γίνει καταγγελίες, τέλος πάντων. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει αποδεκτό. Και το θέμα επίσης του ποια κράτη-μέλη δεν αποδέχτηκαν τι. Ύστερα, χαίρομαι που θίξετε το θέμα της ε, απλούστευσης, ε, της απλοποίησης. Συχνά όμως το αναφέρει το θέμα αυτό το ελεκτικό συνέδριο. Μας είπατε ότι αυτή η απλούστευση αποτελεί σημαντικό θέμα για σας, γιατί πάντα τα ίδια έξοδα, οι ίδιε δαπάνε που είναι περίπλοκες είναι αυτέ που προκαλούν τα προβλήματα και εκνευρισμό και ποσοστό σφαλμάτων. Αλλά είναι περίπλοκα τα πράγματα. Και αυτό με τη σειρά του λοιπόν προκαλεί αγανάκτηση. Σημαντικό ποσοστό του ESF είναι στα απλοποιημένα αυτά, στις απλοποιημένες αυτές τι δαπάνες. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε σε ποια κατεύθυνση κινούμαστε. Για διευκρινίστε μας κάτι γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, επίσης, υπάρχει ένα σύστημα ανταλλαγής γνώσης, ανταλλαγής εμπειριών. Πώς θα συνεχιστεί αυτό το σύστημα. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση υπαριθμών 40, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά εν γέννη ότι η συνεργασία μεταξύ των οργανισμών θα μπορούσε να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω. Φυσικά, αυτό μας οδηγεί στο ερώτημα πώς πρέπει να βελτιωθεί αυτή η συνεργασία, πού υπάρχουν προβλήματα, πού δεν προχωράνε τα πράγματα, πού πιστεύετε ότι υπάρχουν δυνατότητες για καλύτερη συνεργασία και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των οργανισμών. Σε, σε ό,τι αφορά τα προβλήματα μεθοδολογίας τώρα, τι είδους προβλήματα υπήρχαν υπάρχουν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Αρχών Ελέγχου σε ό,τι αφορά την μεθοδολογία. Ή μήπω σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν σκόπιμες και κατάλληλες οι μεθοδολογίες των εθνικών αρχών. Τι προβλήματα παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις εθνικές αρχές ελέγχου. Μήπως υπήρχε και κάποιο πρότυπο, κάποιο μοντέλο Μήπως ε, διακρίνονται κάποια τέτοια μοντέλα σε ό,τι αφορά τα σφάλματα που παρουσιάζονται. Τους τομείς στους οποίους παρουσιάζονται τα σφάλματα. Μήπως υπάρχουν ε, διαφορές σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την αξιοπιστία των εθνικών αρχών. τι δυνατότητε διακρίνεται στο θέμα αυτό. Τελευταία ερώτηση τώρα για το. Για την πρωτοβουλία για τους νέους. Έχουμε με κάποιες πρωτοβουλίες. Στην Γαλλία το ποσοστό απορρόφηση ήταν στο 60%. Σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία. Τι γίνεται στις άλλες χώρες που εφαρμόζουν την πρωτοβουλία για τους νέους. Να απαντήσω για τις ερωτήσεις σας. Σε ό,τι αφορά τις χρηματοοικονομικές ε, διορθώσεις, νομίζω ότι δεν έχουμε προχωρήσει ιδιαίτερως, αν σωστά καταλαβαίνω. Μία διόρθωση έχει γίνει τώρα. Καθαρή διόρθωση και μάλιστα αφορά ένα μικρό ποσό. Πολλά λοιπόν πρέπει να γίνουν ακόμα για τις ε, διορθώσεις ε, αυτές. Κάπου 700.000 δηλαδή αυτή η διορθώση καθαρά. Ναι, αλλά αυτά τα χρονικά διαστήματα μέχρι ότου επιστραφούν τα χρήματα πόσο είναι. Γιατί έχουμε και τον κύριο Μόμπιλε εδώ, το ελεκτικό συνέδριο που πάντα ε, υπάρχουν συζητήσεις για τα ποσά αυτά τα οποία δεν επιστρέφονται ή επιστρέφονται. Και βλέπουμε, δεν πιστώνουμε ότι ε, έχουμε εκκρεμεί 2,7 δις. Το πρόβλημα είναι, δεν είναι ότι τα χρήματα επιστρέφονται αυτόματα. Το πρόβλημα είναι ότι το τμήμα των χρημάτων αυτών μεταφέρεται σε άλλα έργα μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα έργα. Εθνική διόρθωση ή διόρθωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η διόρθωση ανέρχεται σε 2,7 εκατομμύρια. Τα χρήματα αυτά μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα έργα δεν χρειάζεται αυτόματα να επιστραφούν αυτές οι δαπάνες για την περίοδο 2007-2013. Από αυτά τα 2,7 δις, δις έχουν επιστραφεί 73.000. Άρα ο μεγάλος όγκος των δαπανών μεταφέρθηκε σε άλλα έργα, σε άλλα προγράμματα. Δεν έχω επίσης πληροφορίες για το κατά πόσον έχει προσαχθεί σε δικαστήριο οποιαδήποτε, ε, κατά πόσον έχει αποτανθεί σε, στο δικαστήριο οποιαδήποτε κράτος μέλος. Αποδέχτηκαν όλα τα κράτη την ετοιμιγωρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά την απλοποίηση, την απλούστευση, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Να σας το πω και ξεκάθαρα εγώ ως Επίτροπος θα κάνω ό,τι μπορώ για να συνεχίσει αυτή η διαδικασία απλούστευσης. Αυτό είναι προς το συμφέρον και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών και της αποτελεσματικότητας και της Έχουμε θέσει αυτό το στόχο του 50%. Δεν μπορώ να σας πω Πότε θα τον πετύχουμε το στόχο αυτό το συντομότερο δυνατόν. Θα το φροντίσω. Σήμερα το 95% των προγραμμάτων έχουμε απλοποιήσει το 33% των δαπανών. Θα πρέπει το ποσοστό αυτό να αυξηθεί. Θα το κάνουμε αυτά τα επόμενα χρόνια. Ανταλλαγή εμπειριών τώρα. εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο. Να είμαστε σε διαρκή ανταλλαγή με τα κράτη-μέλη, προκειμένου να δούμε αν μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των ταπανών. Θα συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς, θα μιλήσω αγγλικά. Στα αγγλικά τώρα. Πριν το Μάιο του 19 στείλαμε μια επιστολή και τους ε, καλήσαμε να κάνουν ένα πρόγραμμα δράσης για συγκεκριμένα ε, μέσα ε, για το τι θα κάνουν όσον αφορά την υλοποίηση των συστάσεων της αξιολόγησης και οι υπηρεσίες είναι στη διαδικασία του να εκτελέσουν να υλοποιήσουν αυτές τις συστάσεις. Τέσσερις υπηρεσίες έστειλαν στην Επιτροπή το πρόγραμμα δράση, και οπότε δεν προβλέπεται τώρα ε, αναδόμηση της υπηρεσίας και η Γενική Διεύθυνση τη απασχόληση, είπε ότι θα δει τι περιθώριο υπάρχει στο θεσμικό θεσμικό πλαίσιο, τόσο ώστε η αξιολόγηση να μην καλύψει τα μέλλοντα σενάρια και κάποιε μεταβολέ της ε, υπηρεσία, και την αρχιτεκτονική του ή κάποιου συγωνεύσει, γιατί και αυτό αναφέρθηκε ή κάποιε άλλε μεταβολέ τη εντοχή. Και πάει και αυτή, επομένω η καποιου ειδου συγχωνευσει γιατι και αυτο αναφερθηκε η καποιε αλλε μεταβολε τη εντολη και υπαρχει αυτη επομενω η αξιολογηση για κάποιου είδου συμπληρωματικότητε, επικαλύψει για τι υπηρεσίε οπότε να δικαιολογείται, να μείνει όπω είναι τώρα η δομή του και η ανάγκη της ε, αναβαθμισή τους χωρίς συγχωνεύσεις γερμανικά. Όσον αφορά τώρα τα σφάλματα. Uh, yes, ε, audit authorities. Οι ελεγκτικές αρχές χρειάζονται βελτιώσεις ή επισημαίνουν όλα τα λάθη. Όπως γνωρίζετε, έχουν τώρα ένα σύστημα ελέγχου και θεωρούνται αξιόπιστες. Επίσης αναφέρεται το Κωνσταντίνο ότι υπάρχει βελτίωση, υπάρχει αξιοπιστία στο έργο των ελεγκτικών αρχών και θα έπρεπε να γίνουν επαναλήψεις ελέγχων λιγότερες από την πέρση, αλλά έγινε μεγάλη προσπάθεια. Η ΔΕΕ συνεργάζεται συνεχώς με αυτές τις αρχές. Κατευθυντήριες γραμμές, μεθοδολογίες από την Κομισιόν. Κοινή έλεγχη επομένω. Υπήρξε συμφωνία πάνω στα σφάλματα και υπάρχει μια ομάδα εργασίας των ελεγκτών. Και εμείς είμαστε, ο ελληνικό συνέδριο τέλο πάντων είναι παρατηρητής. Και υπήρξε συμφωνία πάνω στα συμπέροντα του ελεγκτικού συνεδρίου και σε σχέση με την τεκμηρίωση. Οπότε η Γενική Διεύθυνση Αποσχόλησης θεωρεί ότι μετά το δικό της έλεγχο μπορεί να στηριχτεί στις ελεγκτικές αρχές για το 75% των λογαριασμών. Τώρα σαν αφορά τα είδη σφαλμάτων. Οι βασικές πήγες σφαλμάτων είναι το ότι σε επιλέξιμες δαπάνες έχει περιληφθεί στις, ε, έχουν περιληφθεί οι δηλώσεις μάλλον στις δαπάνες έχει γίνει παραβίαση των κανόνων σε σχέση με τα εργαλεία της αγοράς και για κάποια μη επιλέξιμα project και δραστηριότητες των ε, ε, επιλέξιμων και είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε αυτές τις αιτίε με συγκεκριμένους ε, τρόπους και να υπάρχει πρόληψη αλλά και διόρθωση και κάποιες ευθύριες γραμμές, κατάρτιση, αναστολές, διακοπές των καταβολών και επίσης διορθώσεις όπου χρειάζονται. Ο φασικός στόχος είναι Πρέπει να συνεχιστεί η στενή συνεργασία με τους ελεγκτές, τόσο ώστε να υλοποιήσουμε τα συμπεράσματα και να δούμε ποια είναι τα εναπομείναντα λάθη για όλα τα προγράμματα και αυτό να είναι κάτω του 2%. Οπότε για να αλλάξει η κατάσταση αυτό που χρειάζεται είναι όπως είπα να γίνουν περαιτέρω απλουστεύσεις ε, στους ε, κανόνες και να ενθαρρύνουμε τις ε, simplified cost options. Τώρα, όσον αφορά την καταπολέμηση της ενεργείας των νέων, έχουμε τα στοιχεία Γαλλίας και Ισπανίας και Ιταλίας. Και μπορούμε να σας δώσουμε στοιχεία και για άλλες χώρες. Δεν τα έχω εδώ, αλλά θα σας τα διαβιβάσω. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και για τα στοιχεία τα οποία θα μας διαβιβάσετε. Και τώρα. Έχουμε τους κοιόδης ηγητές. Συνάδελφα Πλέγκοβα, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Επιτροπή Σμιτ, για την παρουσίαση, για τις εγγραφές ε, απαντήσεις που μας βοήθησαν. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μέρφυ που έκανε τη δική του παρουσίαση είμαι ικανοποιημένη. Έχω μία διευκρίνηση για την ερώτηση 56. Είχαμε ρωτήσει αυτό το οποίο είπατε τώρα τι γίνεται με αυτές τις απλουστευμένες cost options. Και ε, το 2015 είπαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν σε 5 περιπτώσεις για 29 κράτη-μέλη. Και ρωτώ, γιατί καλύπτονται μόνο 20 χώρες και όχι και 28. Μήπως επειδή δεν ενδιαφέρονται τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ε, αυτή την επιλογή αυτές τις, τους τρόπους ή μάλλον ή επειδή κάποιοι δεν είναι προπαρασκευασμένοι να τις εφαρμόσουν σωστά ή πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία η κυρια Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και από πλευρά των Πρασίνων, κύριε Επιτροπέ, που ήρθατε. Thank you for uh, joining our session. Που ήρθατε, έλεγα, στην συνάντηση. Και για να παρελθούμε τώρα σε μια πρωτοβουλία που τη συμμερίζεστε, η πρωτοβουλία για τους νέους και την απασχόληση, αυτό είχε μεγάλη επιτυχία και καταπολεμήθηκε αρκετά σε πολλά κρατημέλη η ανεργία των νέων. Έχουμε στοιχεία για ποιου συμμετέσχουν, για ποιου βρήκανε δουλειά, κατάρτιση, εκπαίδευση και, πέστε μας, έχετε στοιχεία για το ποιοι εγκατέλειψαν αφού συμμετέσχουν στο πρόγραμμα στην πρωτοβουλία να αναπασχόληση τον ένα δεύτερο. Ξέρετε πόσοι ξεκίνησαν την εκπαίδευση και την κατάρτιση και δεν τελείωσαν και τελικά απέκτησαν κάποια δεξιότητα. Και επίση πόσοι αφού αποφύτησαν μετά από έξι μήνες μείναν άνεργοι. Ευχαριστούμε για τα στοιχεία ή για τις απαντήσεις. Χολμαϊερ, σας ευχαριστούμε εμείς. Ο κύριος Κούς είναι ο επόμενος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, παρουσίαση αυτή. Μία ερώτηση έχω να κάνω και γενική φύσεω είναι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προς τον κύριο Επιτροπό Σμιτ. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι στις χώρες που αναφέρατε, στην Ιταλία, στη Γαλλία, αλλά και κυρίως στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και κυρίως στην Ελλάδα, εξακολουθούν να υπάρχει τόσο πολύ υψηλή ανεργία στους νέους, ε, ενώ στη Γερμανία δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι ανάποδα, αντίστροφα σε ό,τι αφορά την απασχόληση και την ανεργία. Πώς το εξηγείτε αυτό το φαινόμενο και τι μπορείτε να κάνετε. Ευχαριστώ. Άλλους δύο βουλευτές, λέει η Πρόεδρος, έχουμε. Σεντόφσκι και Αγγελίκα Βίντσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση και αφορά Euroform, Sendefop, ETF, ε τις, όλες τις υπηρεσίες της απασχολής. Τι γίνεται πλευρά τεχνικής, επιστημονικής, κανονιστικής. Υπάρχουν επικαλύψεις εκεί. είναι γνωστό ότι συνεργαζόμαστε με αυτές τις υπηρεσίες, αλλά μπορούμε να συνεργαστούμε περισσότερο. Και πολλά μπορούν να γίνουν, ούτω ώστε το ETF, το ZITOFOP, το CEDEFOP, το Euroform να συνεργαστούν περισσότερο, να μεταρρυθμιστούν, γιατί θέλουμε να υπάρξει μια τέτοια μεταρρύθμιση γιατί πολλές φορές αυτές οι υπηρεσίες δυσκολεύονται. Και η αποτελεσματικότητά τους δεν είναι τόσο τρομερή. Επίσης, νομίζω ότι στο μέλλον θα είναι δυνατόν να συγχωνεύσουμε δύο-τρεις υπηρεσίες και να έχουμε μόνο μία τελικά ή να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μεταξύ των ε, υπηρεσιών και να έχουν τη διαδικασία πρόσληψης και οι ίδιες διαδικασίες. Και κάποια πράγματα τα κάνουν από κοινό. Για την προβολή δε, τι πιστεύετε. Πιστεύετε ότι είναι προβεβλημένες. Είχα πάει στο Δουβλίνο και τους ρώτησα. Ξέρουν τις υπηρεσίες αυτές του Euroform και αυτές. Γενικά είμαι υπέρ όλων των υπηρεσιών, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε αυτά τα θέματα για την αποτελεσματικότητά τους. Α, επίσης, τι γίνεται με το Ταμείο Αποκοσμιοποίησης και το Καρφούρ. Στο Συμβούλιο δεν έγινε τίποτα. Γιατί αποφάσισε το Συμβούλιο ότι η ψηφιοποίηση δεν είναι πρόβλημα της παγκοσμιοποίησης. Εσείς πώς το βλέπετε. Υπάρχει περίπτωση να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα για το Καρφούρ εδώ στο Βέλγιο και να ξανανοίξει ο διάλογος με το Συμβούλιο. Αγγελικά Βίντσικ. Αγγελικά Βίντσικ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καλώς ορίσατε. Πριν από δύο-τρει εβδομάδε και του προπολογισμού. Point uh, για κάποιο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα για τους νέους. Αυτό είναι αρμοδιότητα κρατών μελών αλλά για τους νέους και για τον προπολογισμό της Ένωσης θα έπρεπε να επενδυθούν περισσότερα στα ε, εκπαιδευτικά συστήματα. Στην Αυστρία έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία των νέων. Είμαι επιχειρηματίας και είμαι υπέρ της μαθητείας όπως έγινε σε Ελβετία, Αυστρία και Γερμανία γιατί και οι τρεις χώρες έχουν χαμηλό δίκτυο ανεργίας. Κύριε Επίτροπε, εσείς τι νομίζετε όσον αφορά το πρόγραμμα για τους νέους. Πώς μπορεί να βελτιθεί στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά το κύριε Επιτροπέ. Τα κράτη-μέλη δεν ε, τήρησαν τους ε, κανόνες τους. Θέλουμε να αλλάξουμε τους κανόνες. Τα πράγματα δυσκολεύουν και στην Επιτροπή ε, προπολογισμού. Είτε έχουμε καθορίσει ως Κοινοβούλιο κάποια κριτήρια μαζί με το Συμβούλιο προφανώς και τα οποία τηρούμε στη συνέχεια Ήταν κάπως εντυπωσιακό αυτό το βήμα. Είτε υπάρχουν οι κανόνες και τους ακολουθούμε, είτε τους αλλάζουμε. Και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόσουμε τους επόμενους ε, κανόνες. Αλλά να μην υπάρχει κανένας κανόνας είναι λίγο περίεργο. Πώς ε, βλέπετε λοιπόν να, εξελίσσονται αυτοί οι κανόνες σε ό,τι αφορά την βιβλία για τους νέους έγιναν κάποιε διαπραγματεύσει, ήταν μαζί και κάποιοι συνάδελφοι και μια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι το πρόγραμμα για την πρωτοβουλία των νέων ε, πήγαινε καλά, αλλά ήταν στον τελευταίο του χρόνο. Δεν έχουμε καταλάβει τελικά τι ισχύει. Και να έλθω και στην ερώτηση της Αγγέλικα Καβίνσικ. Τα φαίνεται τα πράγματα πηγαίνουν καλά στην Ιταλία. Αλλά το θέμα λοιπόν είναι ότι έξι μήνες ποιοι θα είναι θα είναι η κατάσταση γιατί το πρόγραμμα αυτό είναι πλέον ε, δύο χρονών. Τι γίνεται με τους απασχολούμενους, έχουν ακόμα θέση απασχόλησης, έχουν ακόμα δουλειά ή είμαστε πάλι στην αρχή. Αυτό αφορά διαφορετικά προβλήματα που υπάρχουν στην Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες όπου είναι υψηλή ενεργεια <laughs> Πρώτη ερώτηση. Ποια ήταν? Η, τα προστευμένα κόστη. Προωθούμε αυτές τις επιχειρήσεις στα κράτη-μέλη για τα προστευμένα κόστη και όλα τα κράτη-μέλη έχουν πρόσβαση σε αυτή την απλουστευμένη προσέγγιση. Κάποια λίγα κράτη-μέλη δεν, δεν έχουν χρησιμοποιήσει ακόμα αυτή την προσέγγιση, αλλά εμείς ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να τη χρησιμοποιήσουν. Ε, αυτή τη στιγμή καλύπτουν τέσσερις τομείς, εκπαίδευση, ε, κατάρτιση για ανέργου, ε, συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτιση για εκπαιδευτέ. εκπαιδευτές. Με βάση μια μελέτη αυτό το αυτή η απλουστευμένη προσέγγιση δείχνει ότι θα μπορούσε να μειωθεί ε, και το διοικητικό κόστος κατά 25% χάρη σε αυτή τη χρήση των απλουστευμένων ε, ποσών, του απλουστευμένου κόστους. Ε, γι' αυτό ενθαρρύνουν τα κράτη-μέλη να το χρησιμοποιήσουν. Για την ανεργία των νέων. Δεν μπορώ να σας δώσω όλα τα στοιχεία. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τι δεδομένα έχουμε για να σας τα δώσουμε. Αν μετά από έξι μήνες ε, έχουν δουλειά ή όχι, αυτά είναι ειδικά δεδομένα. Ίσως και να υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να το τσεκάρω. Αν τα βρω, τα δεδομένα αυτά, θα σας τα στείλω. Πόσοι εγκαταλείπουν το σύστημα, πόσοι βγαίνουν από το πρόγραμμα. Δεν έχουμε τις πληροφορίες ως πρώην υπουργό Εργασίας που δεν λάμβανε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά που εφάρμοσε αυτή την πρωτοβουλία για τους νέους στο Λουξεμβούργο, έτσι. Είχαμε στο Λουξεμβούργο 20% αποχώρηση από το πρόγραμμα νέων. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία ή σε άλλες χώρες θυμάμαι ότι εμείς είχαμε περίπου 20% των ατόμων που αποχωρούσαν από το πρόγραμμα στο Λουξεμβούργο. Δεν παίρναμε όμω λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η ανεργία των νέων ευτυχώς σε μας ήταν χαμηλότερη από το όριο. Γιατί η ανεργία των νέων είναι χειρότερη σε ορισμένε χώρε και καλύτερη σε άλλε, υπάρχουν πολλοί λόγοι οικονομική, διορθωτική, εκπαιδευτική. Εξάλλου ακούστηκε και μια ερώτηση για το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά υπάρχει και ένας μεγάλος ρόλος, είναι η επαγγελματική κατάρτιση. Κάποιος Αυστριακός το είπε ξεκάθαρα. Νομίζω είστε επιχειρηματίας και το αναφέρατε εσείς. Όταν υπάρχει επαγγελματική κατάρτιση, Παντού η ανεργία των νέων είναι χαμηλότερη αλλά από τις χώρες όπου δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό θέλουμε να πιέσουμε για επέκταση αυτής της επαγγελματική κατάρτισης και υπάρχει και ετοιμότητα και ενδιαφέρον ε, από τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ε, επαρκή επαγγελματική κατάρτιση καθόλου να την ε, εισαγάγουν ή επεκτείνουν. Η επαγγελματική κατάρτιση είναι ένα από τα καλύτερα φάρμακα ένα από τα καλύτερα πράγματα που καταπολεμάται την ανεργία των νέων. Αλλά πρέπει να προσθέσω ότι και το συνολικό οικονομικό πλαίσιο και η ύπαρξη ε, εταιριών που μπορούν να παράσχουν επαγγελματική κατάρτιση είναι και αυτή η σημαντική. Γιατί δεν μπορεί να επιβάλλει την επαγγελματική κατάρτιση στι εταιρείε όταν δεν υπάρχει αυτή η παράδοση. Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε για να προωθήσουμε αυτή την κατάρτιση και στι εταιρείε. Να πείσουμε του επιχειρηματίε. Πάντως αυτό είναι ένα εργαλείο καλό κατά της ανεργίας. Uh, uh, Γιατί η μετάβαση από το σχολείο στην uh, δουλειά, σε μια θέση απασχόλησης, διευκολύνεται. Τώρα για τους οργανισμούς. Έγινε μια μεταρρύθμιση των οργανισμών. Εσείς λέτε ότι είσαστε υπέρ Συγχώνευση κάποιων οργανισμών. Δεν είμαι τόσο πεπισμένο γι' αυτό. Εγώ άρχισα πολύ πρόσφατα να είμαι επίτροπο. Ε, τώρα ανέλαβα τα καθήκοντά μου, αλλά ήμουν σε επαφή με τους οργανισμούς πριν αναλάβω. Και η προστιθέμενη αξία που προσφέρουν οι οργανισμοί για διάφορα θέματα, για διάφορου τομεί πολύ διαφορετικού. Παραδείγματο χάρη το Eurofound, η ΕΚΑ, Οργανισμό χημικών κτλ. Μπορεί να έχουν ε, συνεργασία, αλλά η κάθε μία κάνει και κάτι διαφορετικό και έχει προστιθέμενη αξία η συγκεκριμένη δουλειά τη. Τώρα δουλεύω ε, πάνω σε ένα πολύ σημαντικό θέμα και πολύ διαφορετικό που είναι ε, ο ελάχιστο μισθός και βασίζομαι στην ανάλυση και στα δεδομένα του Eurofound. Έχει κάνει θαυμάσια δουλειά για τους μισθούς και τους ελάχιστους μισθούς στην Ευρώπη. Ε, το έχουμε καλύτερες, το να, για να έχουμε καλές πολιτικές θέλουμε καλά δεδομένα. Γιατί ε- και όταν έχουμε καλά δεδομένα αυξάνεται το αναλυτικό μας δυναμικό. Και το γεγονός ότι ήρθα σε επαφή μαζί με, τις, ε, με τους οργανισμούς αυτούς, με κάνει να λέω ότι ναι, μας δίνουν καλά στοιχεία. Ε, η ΕΚΑ, ας πούμε, με ένα πολύ μικρό προσωπικό, βοηθάει όχι μόνο τους εργαζόμενους για να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας τους και την υγεία και την ασφάλεια, αλλά και τις ίδιες επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρές επιχειρήσεις. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι για τις μικρές επιχειρήσεις μερικές φορές είναι δύσκολο να έχουν και να εφαρμόσουν τα σωστά πρότυπα. Επομένως, θα, θα εγώ θα ήμουν πιο σκεπτικιστής. Δεν θα, δεν θα έλεγα έτσι απλά και εύκολα ότι ναι, μπορούμε να τη συγχωνεύσουμε. Φυσικά πρέπει να προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία και να βελτιώσουμε την ε, λειτουργία τους, να κοιτάξουμε τι κάνουν και αν αυτό που κάνουν επιφέρει προσθέμενη αξία στις πολιτικές μας, για τις πολιτικές μας. Για το επίπεδο γνώσης. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια. Για τον ΕΚΑ, ας πούμε, το παρατήρησε. Γιατί αυτό που κάνουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τι κάνει. Αυτό που κάνει είναι πολύτιμο. Αλλά αρκετά συχνά οι μικρές επιχειρήσεις δεν ξέρουν ποια εργαλεία υπάρχουν και τι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να βελτιωθούν. Μπορούμε λοιπόν να βελτιωθούμε και σε αυτόν τον τομέα της γνώσης. για το ΚΑΦΟΥ, Η Κομισιόν λυπάται όπως και εσείς ε, για την ε, υλοποίηση και εφαρμογή του Ταμείου. Ξέρετε ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός του κανονισμού, θα το επαληθεύσουμε. Και φυσικά πρέπει να προσαρμόσουμε τον κανονισμό και στο μέλλον. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει για να προσαρμόσουμε τον κανονισμό δηλαδή. Τελευταίο ερώτημα. Το τελευταίο το απάντησα εν μέρη. Το να καταπολεμήσουμε την ενεργεία των νέων. Τι σημαίνει. Σημαίνει εν μέρη να διορθώσουμε και τα λάθη του παρελθόντος. Και είναι ποικίλα αυτά τα λάθη. Ας πούμε το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα πρόβλημα συμφωνώ, αλλά είναι εθνική αρμοδιότητα. Είναι πολύ λεπτό θέμα. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα, κοινωνικά, θέματα ένταξης ή ε, μη ένταξης, μετανάστευσης. Όλα αυτά τα θέματα παίζουν το ρόλο τους και οδηγούν σε ανεργία ή μη των νέων. Επίσης, τι γίνεται με τι ανάγκε του. Μερικά παιδιά φεύγουν από το σχολείο, δεν έχουν κατάρτιση, δεν δουλεύουν, δεν είναι σε εκπαίδευση, δεν είναι πουθενά. Θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με του ανθρώπου, να του καλύψουμε. Γιατί αν δεν φτάσουμε σε αυτού, θα είναι προβληματική όλου του η ζωή, αλλά και θα υπάρξουν προβλήματα και για το δικό μας ε, σύστημα. Γιατί θα αναγκαζόμαστε να τους δίνουμε επιδόματα για όλη τους τη ζωή. δεν μπορούμε αυτές τις πολιτικές να τις θεωρήσουμε ως δαπάνες. Είναι επένδυση. Θα έλεγα ότι είναι και επένδυση σταθερότητα των κοινωνιών μας, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Επίτροπε. Και έτσι. Θα ήθελα να δώσω στο τέλος της ε, συνεδρίασης μας το λόγο στο λεκτικό συνέδριο να κάνω και δύο ερωτήσεις και μετά να πάρετε το λόγο για τις απαντήσετε. Το 2005 ε, προσπαθήσαμε να ορίσουμε για το τομέα της απασχόλησης ένα ποσοστό σφάλματος. Θα ήθελα να ξέρω γιατί και πώς έγινε αυτό. Στις συστάσεις επίσης το ελεκτικό συνέδριο μιλά για την απλοποίηση των διαδικασιών και των κανόνων. Την αναφέραμε ήδη. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι τι συγκεκριμένες συστάσεις έχετε να απευθύνετε προς την Επιτροπή για να γίνει αυτή η απλούσταυση. Πού δηλαδή πρέπει να γίνει συγκεκριμένα αυτή η απλοποίηση, αυτή η απλούσταυση. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και πρωτού απαντήσω τις ερωτήσεις σας, να ευχαριστήσω τους βουλευτές και τον Επίτροπο για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την πρωτοβουλία για τους νέους. Ξέρετε ότι ε, έχουμε τρεις ε, ειδικέ εκθέσεις, η τελευταία τον Απρίλιο του 2017 και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα ξαναεμφανιστεί στο πρόγραμμα εργασία. Να επιβεβαιώσει αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ερώτησή σα για την απλοποίηση, κυρία Πρόεδρε. Είδαμε κάποιε περιπτώσει όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει τι εναλλακτικέ απλοποιημένων δαπανών σε ό,τι είπαν, ε, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις άλλους οργανισμούς. Ναι, είναι βασική φορείς πλέον. Αυτή είναι η βασική λοιπόν φορείς και θα πρέπει να γίνει δουλειά εδώ γιατί κάναμε και εντοπίσαμε κάποια ασφάλματα που δεν είχαν εντοπίσει και το ίδιο ισχύει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτοί εντοπίζουν λάθη που δεν υπήρχαν. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι δεν γίνεται τίποτα. Είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Είναι δύσκολο να συντονιστούμε με 28 κρατή-μέλη, με διαφορετικές νοοτροπίες, με διαφορετικά συστήματα. Σε ό,τι αφορά τη δουλειά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, και εδώ είναι πολύ σημαντική η αρμοδιότητά της. Επί του παρόντος ε, επικεντρωνόμαστε στο έργο των άλλων αρχών του χρόνου. Θα κοιτάξουμε καλύτερα τι γίνεται για να έχουμε μια καλύτερη επισκόπηση του συστήματος ελέγχου. Πολλές φορές ε, μου έθεσαν το ερώτημα αυτό, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό σφάλματος για τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Θα ομολογήσω ότι αυτό ήταν πριν από την εποχή μου ως μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου, αλλά ήταν απόφαση ουσιαστικά του Ελεκτικού Συνεδρίου για να υπάρχει τέτοια κατηγοροποίηση ανά κεφάλαιο και όχι για ένα τομέα της πολιτικής. Θεωρούσαν ότι ήταν πιο σκόπιμο να γίνεται τέτοια αξιολόγηση σε περίπτωση, κατά α, επικεφαλίδα και όχι κατά τομέα για την διεύθυνση απασχόλησης και για την διεύθυνση ρίτζιο. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποιο ελάχιστο πώς αριθμό ε, ελέγχων. Και θεωρώ ότι αυτή η περιορισμοί ήταν ένα παράγοντα σε ό,τι αφορά τι συστάσει που κάναμε. Πάντα υποστηρίζαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την εναλλακτική απλοποιημένου κόστου. Το ποσοστό των ε, σφαλμάτων ήταν χαμηλό. Ο λόγος για τον οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε είναι γιατί πετύχαμε το στόχο του 50%, είμαστε στο 23%, ελπίζουμε να αυξηθεί όμως το ποσοστό αυτό. Thank you so much. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ χρήσιμη αυτή ε, παρουσίαση και την έκθεση για τις, ε, ε, τα σχόλια για τη δική μου έκθεση, την οποία θα πρέπει να καταθέσω στις 16 Δεκεμβρίου εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμού. Να ευχαριστήσω και τον Επιτροπό και την ομάδα του. Ίσως θα επανέλθουμε σε κάποια τέτοια θέματα, αλλά όπως και να έχει σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που ήλθατε. So, wir kommen nun zum Περνάμε στο σημείο 10. Ειδική έκθεση υπαριθμών 15-2019 του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου για την εφαρμογή στην Επιτροπή της Δέσμης Μεταρρυθμίσεων του Καθεστώτος των Υπαλλήλων του 2014. Συνεχίζω να μιλάω μέχρι ότου ησυχάσουν τα πράγματα. Μέχρι να δω να φεύγει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητέ κυρία Επίτροπε, να μην είμαι αλλά αν θέλετε να συνεχίσετε έξω προκειμένου να μπορούν οι συνάδελφοι, να μπορέσουν οι συνάδελφοι να ασχοληθούν ε, με την ειδική αυτή έκθεση. Η συγκεκριά μας είναι η Σαμπέλ Καρσιά Μουνιούς και χαίρομαι ιδιαίτερος που έχουμε μαζί μας τον κύριο Πιέτρο Ρούσο, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου. Σας ευχαριστούμε που κάνετε το ταξίδι στις Βρυξέλλες. Να πάρει χάρη λοιπόν το λόγο ο Πιέτρο Ρούσο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Συγκίτρια, κύριοι βουλευτές της Επιτροπής, ευχαριστώ που μας καλέσατε και για το έντονο ενδιαφέρον σας για τον οικονομικό μας έλεγχο και με μεγάλη μου χαρά να σας προς την ειδική έκθεση 15 κάθετος 19 όσον αφορά την εφαρμογή της δέσμης μέτρων του 14 για το προσωπικό. Οι πάλι είναι 60.000 σε θεσμικό όργανα και υπηρεσίες και εδώ συμπεριλαμβάνονται 32.000 εργαζόμενοι πάλι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη χρήση του 2018 οι υποχρεώσεις για το προσωπικό είναι 3,2 δις για την Κομισιόν. Τώρα, όσον αφορά τους ανθρώπους που στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το περισσότερο προσωπικό και άρα το μέτρο κομμάτι του προϋπολογισμού που διατίθεται για το μισθό τους. Θεωρούμε ότι η πιθανή συνέπεια των αλλαγών αυτού του πακέτου μεταρρύθμισης θα είναι παρόμοιο στα θεσμικά όργανα. Όταν είχαμε μεταρρυθμίσει το 2014 στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του προϋπολογισμού για το πλαίσιο 14-20 προέκυψε η πρόταση του Συμβουλίου κάποια επιπλέον μέτρα και δύο ετών καταβολές για τις συντάξεις. Κατόπιν είχαμε περικοπές και κάποιες τροποποίησεις στο καταστατικό του προσωπικού το 14. Πάντα μιλάμε για τη δέσμη μέτρων το 14. Έτσι, εξετάστηκε καλύτερα το τι επηρεάζει τις δαπάνες. Και ε, η ελκυστικότητα των συνθηκών εργασίας. Το βασικό χαρακτηριστικό για τη μεταρρύθμιση ήταν η εξοικονόμηση δαπανών. Επίσης υπήρξε και ανάγκη βελτιώσεων για τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Στον έλεγχο επομένως αυτό εξετάσαμε. Τι γίνεται κατά πόσο αυτά τα μέτρα πέτυχαν το στόχο. Την εξοικονόμηση δηλαδή. Αν βελτιώθηκαν οι ανθρωπινοί πόροι στην Κομισιόν και κατά πόσο υπάρχει εύλογη εποπτεία της ε, εφαρμογής. Καταλήξαμε ότι αυτό το πακέτο του 2014 πέτυχε τις ε, εξοικονομήσεις, τις σκοπούμενες και βελτίωσε και διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Είχαμε κάποιες αρνητικές συνέπειες. Στον αφορά γενικέ διευθύνσει και προσωπικό. Αυτές θα μπορούσαν να έχουν μειωθεί ή να έχουν αποφευθεί νωρίτερα για να ήταν καλύτερα υποπτευόμενοι και προετοιμασμένη αυτή η μεταρρύθμιση. Η δεσμη αυτή του 2014 εξοικονόμησε σημαντικού πόρου. Καλύτερα από όσο περιμέναμε. Και εξοικονόμηση είναι 4,2 δις σε αυτό το πι Και όσον αφορά τις συντάξεις μακροπρόθεσμα έχουμε 19,2 δις. Αυτή η εξοικονόμηση δαπανών για την περίοδο 14-20 όσον αφορά το ΔΕΛΤΑΠΗ είναι ε, το ότι έγινε κάποιο προσωρινό, προσωρινό πάγωμα σε συντάξει και μισθών και επίσης 5% μείωση των, ε, του προσωπικού. Και είχαμε επίσης και κάποια άλλη μεταρρύθμιση της αρρωγής στην ε, καριέρα και επίσης όσον αφορά τις ευκαιρίες για υψηλότερους βαθμούς και για διοικητικούς και για βοηθητικό προσωπικό και πάρα πολλές αυτές τις εξοικονομήσεις για τις διοικητικές δαπάνες που έγιναν να από λιγότερες δαπάνες και στις συντάξεις γιατί υπήρξε αύξηση της ηλικία συνταξιοδότησης και μείωση ε, αντίστοιχης. Οπότε όλα αυτά είναι πλέον των εξοικονομήσεων που ξεκινούν από την μεταρρύθμιση του 2004. Η δέσμη του 2014 όμως έφερε και κάποιες άλλες ε, συνέπειες όσον αφορά τη διαχείριση και η Κομισιόν επίσης ασχολήθηκε με την διαφορετική κατανομή του προσωπικού, ισορροπία ανδρών γυναικών, ε, ηλικιών, αριθμό συμβασιούχων, ε, το φόρτο εργασίας, τον, την ύλη τέλο πάντων των γενικών διευθύνσεων, και την ελκυστικότητα των ε, συνθήκων πρόσληψης, απασχόλησης. Γενικά ήταν ε, τα αποτελέσματα θετικά και αρνητικά. Και έχουμε και δύο σημαντικέ ε, αλλαγέ στην δομή τη σταδιοδρομία που ήδη βοήθησαν τόσο ώστε να υπάρχει περισσότερη σύνδεση αρμοδιοτήτων και μισθού. Οπότε, μακροπρόθεσμα έχουμε αλλαγέ όσον αφορά την κατανομή του προσωπικού ανάλογα με το βαθμό και το μισθό και ε, οπότε το προσωπικό της Κομισιόν έγινε πιο ποικίλο και ανέβηκε το ποσοστό των συμβασιούχων. Αυτή η μεταρρύθμιση οδήγησε σε κάτι φιλικές ρυθμίσεις μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων οπότε υπάρχει τώρα περισσότερη ισορροπία ανδρών και γυναικών 2013 με 2018 παρ' όλα αυτά αυτό δεν οφείλεται στην τροποποίηση του καταστατικού. Θα μειωθεί ανισότητα στους ψηλούς βαθμούς γιατί θα προσλαμβάνονται περισσότερες γυναίκες στους εισαγωγικούς βαθμούς και θα ανεβαίνουν την κλίμακα των ε, η μείωση των προσλήψεων, γιατί έχουμε μείωση του προσωπικού 5% και την, ε, το ανέβασμα της συνταξιωτικής ηλικίας, αυτό βοηθάει στο να υπάρχει μεγαλύτερο προσωπικό σε ηλικία και επίσης ε, και η ηλικία όμως των προσλαμβανομένων ε, συμβάλλει σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, το πακέτο του 2014 έχει και κάποιες αρνητικές συνέπειες για το προσωπικό πολύ σημαντική μείωση της ικανοποίησης του προσωπικού και αύξηση των αναρτικών αδειών. Επιδείνωση στις ε, προσλήψεις όσον αφορά τις αντιπροσωπείες και οι συνθήκες έγιναν χειρότερες για αυτούς που είναι ήδη στο προσωπικό. Λιγότερο ενδιαφέρον για προσλήψεις από τον κόσμο και έτσι ε, ε, ανέβηκαν οι δυσκολίες που υπήρχαν έτσι κι προσωπικά από κάποιες χώρες που ήδη δεν εκπροσωπούνται με πολλούς υπαλλήλους στην Επιτροπή. Επίσης διαπιστώθηκε ότι και τα θετικά και τα αρνητικά της μεταρρύθμισης, εξοικονομήσεις, ε, μείωση της ικανοποίησης και αυτά, αντικατορίζουν το πώς προπαρασκευάστηκε και πώς εποπτεύθηκε αυτή η μεταρρύθμιση. Δεν έγινε αξιολόγηση των ε, πιθανών συνεπειών διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και ποιες ήταν οι συνέπειες των εξοικονομήσεων. Οι ρυθμίσει για την εποπτεία τη Κομισιόν δεν ήταν επαρκεί, ούτω ώστε να επισημανθούν αυτά τα νοικά συμπεράσματα νωρί και σωστά. να σας πω τι συστάσεις διατυπώσαμε μετά από τις παρατηρήσεις μας. Πρώτα πρώτα. Συστήσαμε να υπάρχει ένα πρόγραμμα διαχείρισης του προσωπικού και έτσι όλα να εφαρμόζονται πιο σωστά και να αντιστοιχούν στις ανάγκες. Επίσης να καταρτήσουν ένα πρόγραμμα δράσης για να ελκύσουν έμπειρους από πολλέ εθνικότητε και να τους κρατήσουν. Επίσης, ανακοίνωσε η Κομισιόν το πρόγραμμα για θέματα ανθρωπίνων πόρων για να, αυτό να αντιστοιχεί στην ανάπτυξη του προσωπικού ε, ανάλογα με κάποια δεδομένα και κάποιους ε, δείκτες για να επισημανθεί τι μπορεί να θέσει εν τους στόχους. Επίσης, για το μέλλον πριν γίνει οποιαδήποτε αναθεώρηση του καταστατικού θα πρέπει η Ευρωπαϊκή να επισημάνει τι θέματα πρέπει να καλυφθούν και ποιε θα είναι οι συνέπειε οικονομικέ και μη οικονομικέ σε σχέση με τα μέτρα. Αγαπητοί μου, θέλω να ολοκληρώσω, να ολοκληρώσω ευχαριστώντας ε, το, το επιτελείο μας για τους ε, ελέγχους. Σας ευχαριστώ και ό,τι ερωτήσεις θέλετε προθυμώ να σας απαντήσω. Ευχαριστούμε κύριε Ρούσο. Θα μιλήσω ισπανικά, βάλτε τα ακουστικά σας. Ασκώ και χρέη Προέδρου. Για... Και σας ευχαριστώ ως Πρόεδρος και δίνω και το λόγο στον εαυτό μου, που είμαι και... γιατί είμαι και η συγγήτρια αυτής της έκθεσης. Ως εισηγήτρια λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρούσο για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης και να ευχαριστήσω και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Διορίστηκα πριν από μία εβδομάδα εισηγήτρια αυτής της έκθεσης και επομένως δεν είχα τον απαραίτητο χρόνο για να έρθω σε επαφή με τον κύριο Ρούσο ή με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε με τα συνδικάτα ή με τους εκπροσώπους του προσωπικού δεν έχω τη δυνατότητα να έχω πλήρη εικόνα και να λάβω υπόψη μου την άποψη όλων των ενδιαφερομένων μερών. Τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσω να κάνω όμως κάποιες από αυτές τις συνεδριάσεις και τις επαφές ε, με βάση και τα αποτελέσματα της σημερινής συζήτησης και τις απόψεις των συναδέλφων μου και θα σας ετοιμάσω ε, το συντομότερο δυνατόν ένα έγγραφο εργασία. Ε, το 2014 είχαμε κάποιες διαπραγματεύσεις για τον Πουδουπού 2014-2020. Το πλαίσιο ήταν ότι τα δημοσιονομικά των κρατών μελών υφίστανται φοβερέ πιέσει λόγω τη οικονομική και χρηματοπιστωτική παγκόσμια κρίση. Πολλά από αυτά τα κράτη-μέλη είχαν ανακοινώσει μέτρα για να μειώσουν τι δαπάνε των εθνικών του διοικήσεων και απαιτούνταν και αντίστοιχα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί τα απέτησαν τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούσε να μην το κάνει λοιπόν. Ε, σε εκείνη τη φάση η Κομισιόν δεν έκανε μία αξιολόγηση για τις πιθανές αρνητικές ε, συνέπειες από αυτές τις ε, εξοικονομήσεις. Ούτε μπορούσε να προλάβει και να διορθώσει αυτές τις συνέπειες, τις αρνητικές. Οι μηχανισμοί της Κομισιόν δεν τις επέτρεψαν να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Με βάση τα συμπεράσματα του ελεκτικού συνεδρίου, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, Ειδικά σε αυτή τη φάση τώρα που θα μεταρρυθμίσουμε το καθεστώς των Ευρωπαίων υπαλλήλων, της Ευρωπαϊκής Υπαλληλίας δηλαδή και διαπραγματευόμαστε το νέο ε, πουδουπού, ε, είναι η κατάλληλη ώρα για να ξαναδούμε όλα αυτά τα στοιχεία. Και θα τα δείτε στην έκθεση που θα σας παρουσιάσω στο μέλλον. Θα ήθελα να θέσω μια σειρά από ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινώντας. Ο στόχος του πακέτου μεταρρυθμίσεων ήταν να έχουμε μια πιο αποτελεσματική διοίκηση βασίζεται και να βασίζεται σε δημοσιονομικές περικοπές και να διαχειριζόμαστε καλύτερα τους ανθρώπινους πόρους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Πρώτη ερώτηση. Η ευρωπαϊκή υπαλληλία είναι πιο αποτελεσματική από τότε που έγινε αυτή η μεταρρύθμιση. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και καλύτερα με 5% λιγότερα λιγότερο προσωπικό. Όπως είπε και ο κύριος Ρούσο, εξοικονομήσαμε 4,2 περίπου δις ε, από αυτές τις περικοπές την περίοδο 14-2020, όπως είπε ο κύριος Ρούσο. Πρέπει να, να λάβουμε υπόψη μας την εξοικονόμηση λόγω λιγότερων συντάξεων. Επίσης δεν λαμβάνουμε υπόψη μας το γεγονός ότι έχουμε ε, αναθέσει διάφορες δραστηριότητες ε, προς τα έξω ε, για να διορθώσουμε για να διορθώσουμε την μείωση ας πούμε των ανθρώπινων πόρων. Άρα το κόστος αυτό για, την, για να πληρώσουμε την εξωτερική ανάθεση δεν το υπολογίζουμε αυτό, γιατί αυτό σημαίνει αύξηση. Επίσης ε, γινόμαστε λιγότερο ελκυστικοί, αυξάνονται οι άδειε ασθενεία κτλ. Είναι μερικέ από τι αρνητικέ συνέπειε. Αυτό το εξοικονόμηση του 0,4% αξίζει τον κόπο για όλα τα τις αρνητικές συνέπειες που υπέστη το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, πώς θα αντιμετωπίσετε τη γύραση του προσωπικού. Έχετε ένα σχέδιο προσω... Ε, κομισιόν για να βελτιώσετε τις συνθήκες εργασίας και να ε, είναι ελκυστικό για όλα τα κρατημέλη ε, το να στέλνουν ας πούμε υπαλλήλους ειδικά αυτά που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς. Επίσης, πώς θα λάβετε υπόψη σας την γεωγραφική ισορροπία ή μάλλον την έλλειψη γεωγραφικής ισορροπίας. Το ελεκτικό συνέδριο λέει ότι τον έχουμε συμβασιούχους ε, γίνεται κάτι μόνιμο. Να μην ξεχνάμε ότι τελικά δημιουργούμε μια ευρωπαϊκή υπαλληλία χαμηλού κόστους με αυτούς συμβασιούχους. Και μπορεί αυτό να σημαίνει ότι κάθε έξι χρόνια, ας πούμε, όταν ολοκληρώνεται ας πούμε, η περίοδος αυτών των συμβάσεων, θα πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται. Στο νούμερο 46 παρατηρήσει τη, ε, η Κομισιόν λέει ότι έχουν τη δυνατότητα να παρουσιαστούν σε εσωτερικού διαγωνισμού. Ε, Πόσοι συμβασιούχοι έγιναν ε, υπάλληλοι από το 2014 και μετά με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να μα πείτε, Κομισιόν, σε ό,τι αφορά τι τις άδειε ασθενεία. Συνδέεται αυτό με μέτρα ε, του πακέτου της μεταρρύθμισης όπως ε, ε η μείωση του προσωπικού. Μα είπατε ότι δεν ξέρετε, δεν έχετε δεδομένα για αυτέ τι άδειε ασθενεία. Η Κομισιόν απάντησε στο ε, ελεγκτικό συνέδριο ότι δημιούργησε μία νέα μονάδα ιατρική, καθώ και μία σειρά από ε, εργαλεία εργαλεία πληροφορική, ένα σύστημα προειδοποίηση για να διαχειριστεί τι άδειε ασθενεία και να τι αναλύσει. Πρέπει να μελετήσετε αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στις άδειες ασθενείας και στα μέτρα του πακέτου μεταρρύθμισης. Το κάνατε? Χρησιμοποιείτε αυτή την πληροφορία για να βελτιώσετε τις συνθήκες εργασίας. Θα πρέπει να μας δώσετε αυτά τα δεδομένα, γιατί δεν μας τα έχετε δώσει. Φυσικά να είναι ανώνυμα. Η Κομισιόν με βάση ε, μία μελέτη του 2018 ανάμεσα στο προσωπικό, ε, είπαν, είπε το προσωπικό ότι η ικανοποίησή του βελτιώθηκε σε σχέση με το 2016, αν και το 1 τρίτο του προσωπικού αισθάνεται ότι έχει υπερβολικό φόρτο εργασία. Θα μπορούσατε να μα δώσετε αποτελέσματα αυτή τη έρευνα συνολικά κομισιών ε, βάσει την οποία έχετε καταλήξει κάποια αποτελέσματα. Επίση, στο σημείο 89 ε, μιλάτε για εσωτερικέ στρατηγικέ για να μετριάσετε κάποιε επιπτώσει μεταρρύθμιση. Ποιε ε, είναι αυτέ οι εσωτερικέ στρατηγικέ που χρησιμοποίησατε κομισιόν Και τι αποτελέσματα έχετε πετύχει. Σα ευχαριστώ πολύ, Ιζαμπέλα, για τι πολλέ και πολύ ακριβεί ερωτήσει που μα κάνει. Η συνάδελφό η κυρία Βίντσιχ, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Ρούσο, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, ε, την ειδική αυτή έκθεση και είναι σημαντικό να αναθεωρούμε τις δομές που υπάρχουν. Έχουμε λοιπόν αυτή την ε, μεταρρυθμίση του προσωπικού του 2014, το οποίο είχε ως ε, αποτέλεσμα σημαντικές περικοπές στη χρηματοδότηση. Και είπατε ότι τα κράτη-μέλη μετά την οικονομική κρίση έκαναν περικοπές ό,τι αφορά τα δικά τους έξοδα. Εγώ είμαι νέα βουλευτή και φυσικά αντιμετωπίζω σε διάφορε εκδηλώσει ε, πάντα την κατηγορία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρά τόσο πολλά χρήματα σε προσωπικό και ούτω καθεξής. Αν ήξερα αυτά που ξέρω σήμερα στον προεκλογικό μου αγώνα, θα ήταν πολύ πιο απλό να πείσω κάποιους αντιπάλους και να κατατροπώσω τα επιχειρήματα των ε, πολέμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. πίσω. Θα μπορούσατε να δώσετε λοιπόν ε, εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχει τέτοια αντίκτυπο ε, σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη. Κάτι παρόμοιο είχαμε και για τις κοινέ ε, εταιρείε. Είναι σημαντικός λοιπόν στόχος η ικανοποίηση στον εργασιακό χώρο. Αλλά πιστεύετε ότι τελικά αυτό είχε κάποιο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τη δημοτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί νομίζω ότι πολλοί δεν το ήξεραν καν ότι έγιναν τέτοιε περικοπές. Και τα τελευταία χρόνια η οικονομική κατάσταση έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει δυσκολία πλέον στο να βρει κανείς ε, δουλειά στον δυτικό κλάδο. Και ξέρουμε επίσης ότι η κινητικότητα δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα δεν βλέπω αιτιώδη συνάφεια απαραίτητα μεταξύ των περικοπών αυτών και του γεγονότος ότι είναι λίγο όλο και πιο λίγοι αυτοί που ε, ζητούν δουλειά στα ευρωπαϊκά όργανα. Υπάρχουν επίσης ε, υπάλληλοι από ό,τι ακούμε διοικητικοί για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ε, των περικοπών. Ισχύει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ, Αγγέλικα, λέει η Πρόεδρος. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δώσω το λόγο στον κύριο Κριστιαν Λεβασό για να μα απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν απαντήσω στις ερωτήσεις που τέθηκαν, να πω τρία γρήγορα σχόλια για την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Το πρώτο που κρατήσαμε Είναι θέμα συμμόρφωσης ότι η μεταρρύθμιση του 2014 πρόβλεψε κάποιες διατάξεις που θα οδηγούσαν σε εξοικονόμηση και αυτές οι διατάξεις ε, μεταφράστηκαν σε νομοθετικά κείμενα είτε σε πολιτικές ε, δεσμεύσεις και αυτό που κρατάμε από την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και είναι σημαντικό για την Επιτροπή σας, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σεβάστηκε τις δεσμεύσεις της και τα νομικά κείμενα. Γι' αυτό ακριβώς ε, έκανε αυτές τις περικοπές ε, και προέκυψαν αυτές οι εξοικονομήσεις. Και αυτό που κρατάμε τις περισσότερες παρεμβάσεις σήμερα είναι ότι αυτές οι εξοικονομήσεις συνοδεύτηκαν από μια ε, γκρι κατάσταση ό,τι αφορά τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Ε, πάνω σε αυτό να πω τρία πράγματα. Ένα θετικό πράγμα που τονίστηκε επίσης και από το Επιπτικό Συνέδριο είναι ότι μεταρρύθμιστηκε ε, η δομή της σταδιοδρομίας και υπάρχει καλύτερη σχέση ανάμεσα στο, στο επίπεδο που βρίσκονται ε, και στο βαθμό ε, ευθυνών τους και στον αριθμό των ευθυνών τους. το 2004 η δομή των, των σταδιοδρομιών και ήταν τελείως διαφορετική. Κάτι που είναι λιγότερο θετικό και που εξελίχθηκε σύν το χρόνο είναι αυτό που θα βάλουμε στο κεφάλαιο ευημερία, ας πούμε εντό αγωγικών. Ε, έχετε μια αναφορά σε ό,τι αφορά τις απουσίες, σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση του προσωπικού, όταν έγινε αυτή η έρευνα για την ικανοποίηση του προσωπικού και τα αποτελέσματα που μετρήθηκαν αμέσως μετά τη μεταρρύθμιση του 2014 ήταν ε, χειρότερα από αυτά που είχαμε παρατηρήσει προηγουμένως. Αλλά μετά βελτιώθηκαν στον χρόνο, όταν λήφθησαν κάποια πράγμα, μέτρα από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διορθωθεί το πρόβλημα. Το τελευταίο πράγμα που δεν βελτιώθηκε και που ακούστηκε είναι η γεωγραφική ισορροπία. Και εδώ καταλαβαίνω τις ερωτήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στη σχέση, ε, ανάμεσα στην υποβάθμιση της γεωγραφικής ισορροπίας που συνδέεται με τη μεταρρύθμιση της, ε, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων ε, είναι σημαντικό αυτό για την Κομισιόν και πέρυσι έκανε και δική έκθεση η Κομισιόν για αυτό το θέμα. Είναι το θέμα της ικανότητας της Κομισιόν να προσελκύει υπηκόους από διαφορετικά κράτη-μέλη για να δουλέψουν εδώ στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στην ε, Κομισιόν συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα. Μία τελευταία έκθεση, ε, παρατήρηση για την έκθεση αυτή. Μετά από συστάσεις, μάλλον η Κομισιόν έχει δεχτεί το σύνολο των συστάσεων του ελεγκτικού συνεδρίου. Και φυσικά θα είναι πολύ προσεκτική και θα δώσει συνέχεια στις συστάσεις αυτές. Θα το προσέξει πολύ αυτό το θέμα. Πάω τώρα στα θέματα τα οποία ακούστηκαν. Έχω εδώ τον Διευθυντή της Επιτροπής ε, υπεύθυνο για θέματα υγείας και ευημερία, τον κύριο Ροκ, θα μπορούσε να σα απαντήσει πιο συγκεκριμένα σε ορισμένα ερωτήματα που τέθηκαν. Καταρχά, υπάρχει ένα γενικό ερώτημα. Κατά πόσο είναι ελκυστικά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κατά πόσο είναι αποτελεσματικά επίση. Η μεταρρύθμιση του 2014 μείωσε το προσωπικό και το ενεκτικό συνέδριο είχε ετοιμάσει μια έκθεση ότι που έδειξε ότι η μείωση αυτή του προσωπικού έγινε με βάση τα όσα είχαν προβλεφθεί. Αυτή η μείωση του αριθμού των υπαλλήλων συνοδεύτηκε με αύξηση των συμβαξιούχων. Μάλιστα αυτή τη στιγμή το αναλύει αυτό το φαινόμενο το ελεγκτικό συνεδρίο. Το θέμα που τίθεται είναι να δούμε σε ποιο βαθμό αυτή η επανεξισορρόπηση επηρέασε την ε, ποιότητα των υπηρεσιών. Εδώ το Ενεκτικό Συνέδριο υπογραμμίζει κάποιους κινδύνους που οφείλονται σε αυτή την εξέλιξη. Πρέπει να επανέλθουμε σε ένα ερώτημα που τέθηκε, το θέμα της ελκυστικότητας. Φυσικά, οι συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων είναι πολύ καλύτερες από αυτές των συμβασιούχων. Ε, σε ό,τι αφορά την ελκυστικότητα που έχουμε για τα διάφορα κράτη-μέλη, η Κομισιόν προσελκύει περισσότερο υπαλλήλου ε, στι Βρυξέλλε, εδώ υπαλλήλου στι Βρυξέλλε, από ότι ε, βρίσκει συμβασιούχου, βεβαίω. Είναι σημαντικό αυτό το δούμε. Η σύνθεση του προσωπικού, και αυτή είναι η πρώτη σύσταση του, ε, του ελεκτικού συνεδρίου, παίζει μεγάλο ρόλο στο κόστος, στη διαχείριση της γνώσης στην διαιώνιση της ευρωπαϊκής υπαλληλία και στην ικανότητά μας να προσελκύσουμε προσωπικό. Φυσικά πιο εύκολα θα γεμίσουμε μόνιμες θέσεις υπαλλήλων παρά ε, συμβασιούχων. Φυσικά, είπατε ότι θα πρέπει να δούμε μεθοδολογικά το πώς δουλεύει η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχει γεωγραφική εξισορρόπηση, δεν υπάρχει διαφορετική μεθοδολογία. Απλώ μετρήσαμε διαφορετικά πράγματα εμεί και το ελεκτικό συνέδριο. Αλλά συμφωνούμε με τα νούμερα, γιατί χρησιμοποιούμε τα ίδια νούμερα. Απλώ πήραμε. Ε, είδαμε το ίδιο φαινόμενο από άλλη σκοπιά. Μετρήσαμε άλλε παραμέτρου δηλαδή. Τα συμπεράσματά μα όμω είναι πολύ παρόμοια. Χρησιμοποιούμε τα ίδια πράγματα. Τα ίδια νούμερα. Εμεί ω Κομισιόν ε, είδαμε από πού ξεκινάει ένας διοικητικός υπάλληλος, από ποιο βήμα ας πούμε, έτσι. Και αυτή είναι η βάση ε, για την ευρω... μελλοντική ευρωπαϊκή ε, υπαλληλία. Όταν κοιτάμε τα νούμερα του ελεκτικού συνεδρίου, ε, ε, στην πραγματικότητα στο ίδιο καταλήγουμε, με άλλες παραμέτρους όμως το μετράμε. Τώρα, γι' αυτό που συνέβη το 2014, οι συμβασιούχοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε εσωτερικούς διαγωνισμούς αυτή η δυνατότητα υπήρχε στο παρελθόν για τους έκτακτους υπαλλήλους. Υπήρχε πάντα, αλλά για τους συμβασιούχους ε, ξεκίνησε μόνο από το 14, 14 και μετά. Έκτοτε δύο διαγωνισμοί για την Κομισιόν έγιναν για τους συμβασιούχους, ένας α, διαγωνισμός το 2016 και ένας άλλος το 2018. Αυτή η διαγωνισμοί ήταν ανοιχτοί και στου ε, έκτακτου υπαλλήλου και στου ε, μόνιμου υπαλλήλου. Στο διαγωνισμό του 2018 είχαμε πάνω από 6.000 ε, υποψηφίου που συμμετείχαν σε εσωτερικού διαγωνισμού και μεταξύ αυτών χίλιοι περίπου συμβασιούχοι είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αυτόν τον εσωτερικό διαγωνισμό για να γίνουν μόνιμοι υπάλληλοι. Σε ό,τι αφορά το σύνορο των ερωτήσεων για την ευημερία και την υγεία των υπαλλήλων θα δώσω το λόγο στον Χριστιαν Ρόκα, που είναι διευθυντής υπεύθυνο για αυτά τα θέματα στη Γενική Διεύθυνση, αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Βεβαίω, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ρόκ, λοιπόν. Παρά αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι σχετικά σύντομος. Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του 2014 η Επιτροπή ευθύς αμέσως έλαβε ε, τα, μέτρα για να δει πώς είναι η κατάσταση για αυτή την μεταρρύθμιση και στην αρχή είχαμε ε, μια μελέτη για, την, για τις αρχές 14-15 για να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα, τα ενδεχόμενα τα οποία θα μπορούσαν αρνητικά όσον αφορά τις καλεστικές εργασίες και όσον αφορά τους εργαζόμενους τις επιπτώσεις στην υγεία. Αυτό το οποίο είπε η συγγήτρια. Είχαμε μια ειδική μονάδα που παρακολουθεί τις αρνητικές άδειε, όχι, όχι ελεγκτικά, αλλά για να διαχειριστούμε, να παρακολουθήσουμε τι γίνεται με τους συναδέλφους και ο στόχος είναι να βοηθήσουμε την επιστροφή στην εργασία στις καλύτερες συνθήκες με της έκθεσης. Χαράξαμε μια φιλόδοξη Fit at work. Σε φόρμα στη δουλειά με έξι πυλώνες, έξι άξονες και ο στόχος είναι διάφορες δραστηριότητες. Σωματική, πνευματική υγεία, ένταξη στην ε, κοινωνική ζωή, στα κράτη-μέλη που φιλοξενούν τα θεσμικά όργανα και γενικότερα για τις εργασιακές σχέσεις. Μάλλον για τις σχέσεις στην δουλειά, στον χώρο της δουλειάς, το, χώρου, τους χώρους, τα γραφεία και άλλα. Έτσι ξεκίνησαν προσπάθειες από πολλές υπηρεσίες της Κομισιόν. Και προσπαθήσαμε να υπάρξει καλή διάθεση και αρκετή επιτυχία σημειώθηκε και μετά κάναμε κάποια γκάλωπ στο προσωπικό το 2015 ήταν αρνητικέ οι όσον αφορά την κατάσταση και την αντίληψη των συνθήκων τη δουλειά και το τι κάνει η Κομισιόν για του υπαλλήλου. Πέρασαν δύο χρόνια και είδαμε ότι κατά 20 πόντου είχε αυξηθεί η ικανοποίηση των συναδέλφων. Δεν θα πρέπει να πετάμε τη χαρά μα. Θέλουμε να περάσουμε το 50% και ήμασταν 30 μόνο και πήγαμε 50 και έτσι συνεχίζουμε την πρωτοβουλία και ελπίζω θα πάμε ακόμα καλύτερα. Με λίγα λόγια, είδαμε ποια είναι, είναι, ποιοι είναι οι κίνδυνοι ψυχοκοινωνικοί σε όλες τις γενικές διευθύνσεις και παρακολουθούμε, υποπτεύουμε να δούμε τι γίνεται και από πλευράς νομικής κάλυψης για την παρενόχληση και βλέπουμε τι γίνεται και αλλάζουμε αν χρειαστεί το χρόνο εργασίας. Βλέπουμε τι γίνεται σε σχέση και με τον ε, κανονισμό υπηρεσιακή κατάστασης, τι γίνεται με τους αναπήρους ή μέλη τη οικογένεια που έχουν αναπηρία. Και συνέχεια κοιτούμε τι γίνεται με την νομική βάση στην Κομισιόν για να βελτιωθεί η κατάσταση ένα σωρό αθλητικές δραστηριότητε, ε, δίνονται κίνητρα στο προσωπικό. Όλα αυτά τα έχουμε. Και είναι στη διάθεσή σας, αν τα θέλετε, στο Κοινοβουλίο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή επισκόπηση σε ό,τι αφορά τις ε, αποφάσεις αυτές και σε ό,τι αφορά τους προσωρινούς ε, εργαζομένους και τους ε, συμβασιούχους και τους συμβούλους. Και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω την εισηγητρία κατά πόσον έχει οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή κάποια επιθυμία ή κάποια παρατηρήση όχι. Να δώσω λοιπόν και πάλι το λόγο στον κύριο Ρούσο για να τοποθετηθεί. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Να σας πω πρώτα-πρώτα. Εννοείται ότι το θέμα είναι περίπλοκο. Ε, το θέμα είναι η προπαρασκευή, τα μέτρα, αυτό το οποίο συζητούμε και υπάρχουν πολλές μεταβλητές. Θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτά η Επιτροπή. Δεν γίνεται πάντα αυτό, δεν υπάρχει πάντα ο έλεγχος. Πολύ καλά τα είπε η εισηγήτρια. Έγινε αυτή η μεταρρύθμιση σε μια συγκυρία κρίσης σε όλη την Ευρώπη. Είχε ήδη ξεκινήσει λίγο χρόνια πριν και συνεχιζόταν. Και υπήρχε πίεση στα κρατημέλη για να μειώσουν τις ε, δαπάνες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τελικά έγινε, έγινε ξεγνώμηση δαπανών και μέσα στα ίδια τα κράτη-μέλη. Βέβαια, υπάρχει εδώ το πολιτικό στοιχείο, αλλά δεν είναι δουλειά μου να ασχοληθώ με αυτό. Οικονομικός ελεγκτής είμαι. Οπότε δεν μπορώ να σχολιάζω αυτούς που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Οπότε είπαμε ότι αυτή ήταν η πολιτική τάση να μειωθούν οι δαπάνες πάγωμα μισθών, συντάξεων για κάποιο διάστημα. Παράλληλα είχαμε μια διοργανική συμφωνία. Μείωση 5% του προσωπικού. Για όλα τα θεσμικά όργανα. Αλλά λόγω μεγέθους αυτό αφορούσε κυρίως την Κομισιόν. Οπότε πρέπει να συμμορφωθεί και στη νομοθεσία της η Κομισιόν. Οπότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθετεί η Κομισιόν επομένως οι παρατηρήσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεσή μας έγιναν αποδεκτές από την ε, Κομισιόν. Ισχύουν αυτά που είπαμε. Ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός, καλύτερη αξιολόγηση εκ των προτέρων για τις συνέπειες εκείνων των μέτρων εξοικονόμησης δαπανών. και στη συνέχεια να υπήρχε εποπτεία, παρακολούθηση της εξέλιξης κλπ. Μπορώ μπορούμε να πούμε για την έκθεση ότι έγινε κάποια συλλογή στοιχείων με αντικειμενικότητα δεν υπήρξε κάποια ένσταση από την Κομισιόν για αυτά τα στοιχεία. Θεωρήθηκε ότι αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Οπότε, συμφωνήσαμε επί των συμπερασμάτων. Αναμενόμενες οι εξοικονομήσεις και με το παραπάνω. Μεγάλο τμήμα της ήταν από, από το πάγωμα των μισθών. Βέβαια, εκ των υστέρων έκρινε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι ήταν παράνομο το πάγωμα των μισθών. Έτσι έγινε η οικονομία. Επίσης, με τις μεταρρυθμίσεις για την σταδιοδρομία έχουμε πιο μακρόπνοες ε, οικονομίες λόγω των ρυθμίσεων για μισθούς και συντάξεις. Επομένως, δεν λέμε ότι υπάρχει αυθαιρεσία γιατί αν ήταν, κρίθηκε ότι ήταν ε, αναγκαία η οικονομία και αν εντό εισαγωγικών αυτό επιβλήθηκε από τα κέντρα των πολιτικών αποφάσεων θα έπρεπε όμως να ληφθούν υπόψη οι αρνητικέ συνέπειες που δεν έλειπαν. Και μια που τα είπε πολύ καλά η κυρία Γκαρθία, τα είπε καλά και διεξοδικά, να μην επανέλθω σε αυτό. Αυτό για τις αρνητικές συνέπειες της μεταρρύθμισης. Άρα θα πρέπει να αντιλήσουμε κάποια συμπεράσματα, να πάρουμε μαθήματα από το τι έγινε, όπως το αναγνωρίζει η Κομισιόν και θεωρώ ότι οι σχετικές προτάσεις πάνε στη σωστή κατεύθυνση, όλα αυτά να λεφθούν υπόψη και να γίνει προσπάθεια για τα πιο ενδεδειγμένα μέτρα. Βράχει πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Και έτσι να απαλληλθούν οι αρνητικές συνέπειες. Νομίζω ήταν χρήσιμη η έκθεση. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε στην καλύτερη διαχείριση. Είδε εφαρμοστές διατάξεις όπως τα είπε και η συγκίτρια, θα συζητηθούν στις ε, διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αντίθετα σήμερα το πρωί καταφέραμε να τελειώσουμε και λίγο πιο νωρίς. Ε. Να ευχαριστήσω όλους σας ε, που είναι εδώ από σήμερα το πρωί που συμμετείχαν σε όλα αυτά τα σημεία τη ημερήσια διάταξη. Να ευχαριστήσω το λεκτικό συνάδριο, τον κύριο Ρούσο, όλο ιδιαίτερο. Και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ευχαριστήσω για τι πληροφορίε που μα ε, υποσχέθηκε. Και σας εύχομαι καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο.